θεία τους και παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Με την πεποίθηση αυτή λοιπόν θα πω πρώτα ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη που έλαβε τελική μορφή η έκθεση και μπορούμε τώρα να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες διότι νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία της εργασίας μας επί της ε, πολιτικής συνοχής ήταν κάτω από αυτό το μεγάλο, το μεγάλο νέφος της ε, δημογραφικής εξέλιξης και ε, βεβαίω αυτά τα έχουμε λάβει υπόψη μας μέχρι τώρα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική η ε, συγκεκριμένη μελέτη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στους εμπειρογνώμονες και νομίζω ότι θα αρχίσουμε με την κυρία Σάμεκ Λοντοβίτσι, μετά ο κύριος Κάρλος και μετά θα ακολουθήσουν και άλλοι. Ε, ο τελευταίος μάλλον εμπειρογνώμων. Άρα λοιπόν ας ακούσουμε πρώτα την κυρία Σάμεκ Λοντοβίτσι. Η κυρία Σάμεκ Λοντοβίτσι, ευχαριστώ που μας καλέσατε να που μας προσκαλέσατε να, εξετα... να ε, παρουσιάσουμε τη μελέτη που είναι ε, μεγάλη και το πρώτο κομμάτι είναι βέβαια η συγκριτική μελέτη και το άλλο το βαρύ κομμάτι της μελέτης είναι οι δέκα μελέτες που, οι 10 έρευνες που λάβαμε υπόψη. Τώρα, λίγα λόγια για τον στόχο και το περιεχόμενο της μελέτης. Ο στόχος ήταν να κάνουμε μια επισκόπηση των περιφερειακών δημογραφικών δομών και τάσεων και να δούμε ποιος υπήρξε ο ρόλος της πολιτικής συνοχής ή των πολιτικών συνοχής στα έτη 2007 έως 2013 στην περίοδο προγραμματισμού δηλαδή των ετών αυτών για να δούμε τι είδους ενδείξεις μπορούμε να συναγάγουμε από το προγραμματισμό αυτό για να δούμε τι θα γίνει για την επόμενη περίοδο. Εξετάσαμε λοιπόν τη σχετική τεκμηρίωση και τα δεδομένα για δημογραφικές και εδαφικές τάσεις. Επανεξετάσαμε την ε, προγραμματική περίοδο 2007-2013 με εξετάζοντας σχετικά έγγραφα και εξετάσαμε τα έγγραφα προγραμματισμού καθώς και τα δημοσιονομικά δελτία για να δούμε δηλαδή ποια κονδύλια κατευθύνθηκαν προς μέτρα τα οποία έχουν σχέση με τις δημογραφικές αλλαγές. Και κάναμε και σε βάθος ανάλυση πεδίου με έξτρα συλλογή δεδομένων σε 10 περιφερειακές μελέτες, case studies, που λάβαναν ε, υπόψη χαρακτηριστικές κοινωνικο-οικονομικές και δημογραφικές συνθήκες. Και τέλος έχουμε και ορισμένα συμπεράσματα και επιπτώσεις για την πολιτική για την περίοδο 2014 έως 20. Τώρα για τα βασικά δημογραφικά, βασικές μάλλον δημογραφικές και εδαφικές τάσεις, εκεί θα είμαι αρκετά σύντομη γιατί θα μιλήσουν για αυτά και άλλοι. Είδαμε ότι η βασική πρόκληση για την περιοχή της Ένωσης είναι η γύρανση του πληθυσμού αναμένουμε μείωση του πληθυσμού και λόγω γύρανσης και λόγω μείωσης της γεννητικότητας. Το μέγα πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μείωση του ε, πληθυσμού που βρίσκεται σε ε, ηλικία ικανότητας προσεργασία. Λιγότεροι άνθρωποι λοιπόν θα είναι, σε, είναι και θα είναι σε ηλικία που μπορούν να δουλέψουν και, να, και αναγκάζονται να στηρίξουν μεγαλύτερο αριθμό ηλικιωμένων ανθρώπων. Άρα οι προκλήσεις αυτές είναι σημαντικές και έχουν και πολύ ισχυρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που θα σας εξηγήσω αργότερα. Οι διεθνείς μεταναστεύσεις και γενικότερα στην Ευρώπη είναι ωστόσο και η σημαντική όθηση για τις αλλαγές του πληθυσμού. Παραπάνω από τρία τέταρτα των αυξήσεων του πληθυσμού ήταν από καθαρές εισόδους μεταναστών ακόμα και αν υπάρχουν βέβαια αυτές οι γενικές τάσεις σε όλη την Ευρώπη έχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Υπάρχει μεγάλη ετερογένεια μεταξύ των περιφερειών. Ορισμένες περιφέρειες βλέπουν να μεγαλώνει ο πληθυσμός τους, αλλού μειώνεται. Ορισμένες περιφέρειες έχουν σημαντικές εισόδους μεταναστευτικών ρευμάτων, άλλες, ιδίω από τις νοτιοανατολικές χώρες, βλέπουν τον κόσμο να φεύγει για να πηγαίνει να βρει δουλειές σε άλλες χώρες. Επίσης, μεγάλες διαφορές σημειώνονται και εντός των ίδιων των περιφερειών όσον αφορά τη νέα εδαφική κατανομή των ομάδων πληθυσμού. Για παράδειγμα, στα αστικά κέντρα Αυξάνεται ο πληθυσμός στις πρωτεύουσες, σε, ορισμένα αστικά κέντρα ο κόσμος φεύγει από το κέντρο και πηγαίνει στις περιφέρειες των ε, αστικών κέντρων, ιδίω νεότερες νέες οικογένειες με μικρά παιδιά, ενώ στο κέντρο των πόλεων παραμένουν κυρίως ηλικιωμένοι και μετανάστες. Υπάρχουν επίσης ορισμένες, μάλλον μικρότερες πόλεις που βλέπουν να μειώνεται ο πληθυσμός τους, ιδίως δε στην Ανατολική Ευρώπη και σε ορισμένες περιφέρειες της Δυτικής Ευρώπης. Το ίδιο υπάρχει πρόβλημα των περιοχών της Υπέθρου, οι ορεινών περιοχών, που επίσης βλέπουν να μειώνεται ο πληθυσμός τους και ο κόσμος που μένει εκεί είναι ε, περισσότερο απομονωμένος. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι μεγάλες διαφορές που απαιτούν πολιτικές που να είναι βασισμένες σε ξεχωριστές προσεγγίσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση, διότι οι διαφορές μέσα στην ίδια χώρα αλλά και μεταξύ περιφερειών και εντός των περιφερειών είναι τόσο μεγάλες που χρειαζόμαστε ειδικέ πολιτικές στοχευμένες στις ε, ε, τοπικές συνθήκες. Δεν ξέρω αν βλέπετε καθαρά την διαφάνεια στην οθόνη. Βλέπετε Ωστόσο, εκτιμήσεις, δημογραφικές προβλέψεις για τις ε, περιφέρειες των, της Ευρώπης των 27 για τα έτη 2008-2030. Οι ανοιχτές γαλάζιες περιοχές είναι οι περιοχές όπου πιθανότατα θα υπάρξει αύξηση του πληθυσμού. Είτε λόγω θετικών φυσικών τάσεων, είτε λόγω εσωτερικής μετανάστευσης η οποία αντισταθμίζει την ε, μείωση των εθνικών πληθυσμών. Οι σκούρες κιανές περιοχές είναι περιοχές όπου θα είναι πιθανότερο να σημειωθεί μείωση του πληθυσμού. Είτε λόγω μείωσης της φυσικής αύξησης, είτε λόγω μετακίνησης προς τα έξω ε, των πληθυσμών από λοιπόν, τα στοιχεία αυτά μπορείτε να δείτε ότι η αύξηση πληθυσμού αναμένεται ιδίω στα δυτικά και βόρεια. Μείωση των πληθυσμών βλέπετε ιδίω στην Πολωνία και στην κεντρική Ευρώπη καθώς και στις χώρες της Βαλτικής και τις Ανατολικές χώρες ενώ η Νότια Ευρώπη έχει ορισμένες περιοχές όπου θα αυξηθεί ο πληθυσμός και άλλες όπου αναμένεται να μειωθεί. Λοιπόν είναι πάρα πολύ διαφοροποιημένη η εικόνα. Όπως ανέμενα και από πριν, οι δημογραφικές αυτές τάσεις έχουν σημαντικές επιπτώσεις και σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη και σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή. Για αυτές τις κοινωνικονομικές επιπτώσεις το μέγα πρόβλημα είναι η μείωση του πληθυσμού που βρίσκεται σε ηλικία όπου μπορεί να εργαστεί. Αν λοιπόν δεν υπάρξουν ειδικέ πολιτικές που να ενισχύσουν το τμήμα αυτό του πληθυσμού, σημαίνει τότε χαμηλότερη παραγωγικότητα και λιγότερη ανάπτυξη, γιατί λιγότερος κόσμος θα δουλεύει. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν το πρόβλημα αυτό, χρειάζεται να αυξήσουμε το ρυθμό συμμετοχής το ποσοστό συμμετοχή ιδίω γυναικών και ηλικιωμένων. Χρειάζεται επίσης να βελτιώσουμε τις συνθήκες της αγοράς εργασίας και πρόσληψης μεταναστών που έρχονται σε αυτές τις χώρες. Όσον αφορά τώρα τις κοινωνικές επιπτώσεις, το πρόβλημα είναι η απομόνωση και ο κίνδυνος να πέσουν σε επίπεδα φτώχειας μεγάλες πληθυσμικές ομάδες, ιδίως ηλικιωμένοι που ζουν, που ζουν μόνοι τους, άνθρωποι που ζουν σε περιοχές της Υπέθρου, οι ε, ορεινές περιοχές, ή άλλες απομονωμένες περιοχές, επίσης μετανάστες και αυτό σημαίνει επίσης αύξηση κόστους για τους δημόσιους προϋπολογισμούς σε ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία, δαπάνες για συντάξεις, επίσης για τις ιατροφαρμακευτικές ε, περιθάλψεις και αυτά όλα τα κόστη θα αυξηθούν. Υπάρχει λοιπόν, τίθεται λοιπόν πρόβλημα βιωσιμότητας του κοινωνικού κράτους λόγω της τάσης γύρανσης του πληθυσμού. Υπάρχουν λοιπόν επιπτώσεις σε πολλούς τομείς πολιτικής από τις αλλαγές αυτές, τις δημογραφικές αυτές αλλαγές. Ξεκινούμε από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας μέχρι, τις, ε, μέχρι τη βιομηχανική πολιτική, την πολιτική απασχόλησης, για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που προέρχονται από την τάση αυτή, χρειαζόμαστε περισσότεροι άνθρωποι να μπουν στην αγορά απασχόλησης. Χρειαζόμαστε λοιπόν πολιτικές απασχόλησης, χρειαζόμαστε νέες επιχειρήσεις, νέες εταιρείε που να ε, τονώσουν την παραγωγή, άρα βιομηχανικές πολιτικές. Χρειαζόμαστε πολιτικές για την ε, χωροτακτική ρύθμιση και των αστικών κέντρων και της υπέρθου. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια να μειωθούν αυτές οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις αστικές περιοχές και στις, χω... στις περιοχές της υπέρθου, πρωτεύουσες και πόλεις δορυφόρους κλπ. Χρειαζόμαστε και υποδομή η οποία θα εξασφαλίσει τις ε, μετακινήσεις μεταξύ των περιοχών για να αποφευθεί απομόνωση. Άρα και μεταφορές, συγκοινωνίες δηλαδή, αλλά και τεχνολογία επικοινωνιών. Επίσης χρειάζεται μια κοινωνική υποδομή, η δημιουργία δομών υγείας, παιδείας και ούτω Χρειάζεται επίσης ισότητα φύλων καθώς και οικογενειακές πολιτικές για να τονώσουμε την γονιμότητα και να στηρίξουμε τις γυναίκες ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εργασία απασχόλησης. Εφόσον οι γυναίκες μπουν περισσότερο στην αγορά εργασίας θα μπορέσουν να εξισορροπήσουν κάπως τουλάχιστον τις αρνητικές επιπτώσεις της ε, γύρανσης του πληθυσμού. Χρειαζόμαστε επίσης πολιτικές εκπαιδεύσεως, καταρτήσεως και για τους νέους αλλά και για τους ηλικιωμένους. Χρειαζόμαστε βεβαίως πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης των μεταναστών. Όλες αυτές οι πολιτικές έχουν ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση των δημογραφικών τάσεων. Το ίδιο σημαντικό είναι να συνεργαστούν οι διάφοροι θεσμοί. Χρειαζόμαστε δηλαδή παρέμβαση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Περιφερειών, όργανα τα οποία ήδη έχουν κάνει πολλή δουλειά, διότι άρχισαν ήδη από το 2005 να θέτουν τα θέματα αυτά στις ατζέντε τους, ε, προσφέρουν κίνητρα για συζητήσεις, για παραγωγή δεδομένων. Έχουμε πολλούς δείκτες τώρα και δεδομένα που είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα προβλήματα στο τοπικό επίπεδο. Έχει δοθεί προσοχή στην νομοθετική ρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων στον κανονισμό του 2007 της προγραμματικής περίοδου 2007 έως 2013 περιλαμβάνεται και άρθρο για τα διαρθρωτικά ταμεία τα οποία καλούνται να ασχοληθούν με τις δημογραφικές εξελίξεις. Και επίσης για τον Ρίτο 2020 περιλαμβάνεται ο στόχος η αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών. Μεταξύ αυτών των προκλήσεων δηλαδή περιλαμβάνεται και αυτό. Καθώς επίσης στις εμβληματικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται ειδικέ ενδείξεις για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της γύρανσης, επίσης για διαβίου κατάρτιση, για θέματα άλλα σχετικά. Επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προ οκταετίας περίπου άρχισε να συζητεί τα θέματα αυτά και έχετε το ψήφισμα του 2011 για τις επιπτώσεις των δημογραφικών πολιτικών στο περιφερειακό επίπεδο που είναι πραγματικά εξαιρετικά επίκαιρο. Εμείς διαπιστώσαμε ότι τα αποτελέσματα, τα πορίσματα μάλλον της μελέτης είναι πολύ συνεκτικά με το περιεχόμενο του ψηφίσματός σας. Και επίσης οι επιπτώσεις της πολιτικής είναι πολύ ε, συνεκτικές με το ψήφισμα. Στο επίπεδο των χωρών μελών αυτά που έχουν γίνει είναι κυρίως οι αναθεωρήσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων και των συστημάτων υγείας. Με πρόβλημα κυρίως βέβαια την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων αδαπανών για τις συντάξεις και την υγεία. Με τη σκέψη κυρίως να μειώσουν όσο το δυνατόν τις δαπάνες για να αποφευθεί στο μέλλον μια εκτόξευση των δημοσίων δαπανών στους ε, τομείς αυτούς. Αρχίζει σιγά σιγά και ε, το active aging να παίζει ένα ρόλο. Έχει δοθεί δε ιδιαίτερη προσοχή στις δαπάνες της πολιτικής συνοχής. Όχι πάντα ρητά, όμως ορισμένα από τα θέματα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί και από την πολιτική συνοχή στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδα. Ο ρόλος της πολιτικής της συνοχής λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικός, ιδίως για τις περιφερειακές και τοπικές πολιτικές και ιδίως διότι τα περισσότερα σημαντικά θέματα του Περιφερειακού και του Κοινωνικού Ταμείου μπορούν να αντιμετωπίσουν δημογραφικούς κινδύνους αφού έχουν σχέση με θέματα που και αυτά με τη σειρά του σχετίζονται με τις δημογραφικές αλλαγές. Εμείς έχουμε ταξινομήσει τις προτεραιότητες αυτές των θεμάτων και διαπιστώσαμε εξετάζοντας τα ποσά των δημοσιονομικών πόρων που κατευθύνθηκαν προς τα εκεί ότι 19% του περιφερειακού, κοινωνικού και ταμείου συνοχής έχουν διατεθεί για προτεραιότητες που άμεσα ή έμεσα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των δημογραφικών αλλαγών. Άρα έχουν γίνει πολλά πράγματα ήδη, ακόμη και αν Δεν μνημονεύονται ρητά τα θέματα αυτά μεταξύ των ε, οριζοντίων αρχών. Εδώ ε, επίσης στη διαφάνεια αυτή βλέπετε πώς κατανεμήθηκαν οι πόροι στις διάφορες ε, περιφέρειες των ταμείων που προανέφερα. Σε μέτρα δηλαδή τα οποία έχουν σχέση με την δημογραφική αλλαγή. Οι σκούρες και νέες περιοχές είδαν να διατίθεται σε αυτές τα περισσότερα και μεγαλύτερα κονδύλια από τους πόρους αυτούς. Οι ανοιχτές και ανές ε, περιοχές έχουν λάβει λιγότερα κονδύλια. Και θα δούμε τώρα και τι είδους μέτρα έχουν χρηματοδοτηθεί ε, από το Ταμείο της ε, Πολιτικής Συνοχής. Με το Περιφερειακό Ταμείο, Περιφερειακής Αναπτύξεως δηλαδή, Εκεί οι δαπάνες είχαν σχέση κυρίως με την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών, υγεία, εκπαίδευση, κοινωνικές υποδομές για την αναζωογόνηση αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου. Εκεί ήταν κυρίως οι δύο περιοχές παρέμβασης σημαντικές για τη δημογραφική αλλαγή. Επίσης το Διαρθρωτικό Περιφερειακό Ταμείο χρηματοδότησε και έρευνες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον γυράσκοντα πληθυσμό. Νέοι τομείς αυτοί τεχνολογικής ε, εξέλιξης που μπορεί να είναι πολύ σημαντικές και που θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τα μέτρα που λαμβάνονται για να μπορούν να απασχολούνται περισσότερο οι ηλικιωμένοι, active aging δηλαδή, ε, ενεργός γύρανση, στήριξη των γυναικών επίσης για να βρουν δουλειά, επίσης για τους νέους και για τους μετανάστες. Αυτές ήταν οι ομάδες στόχοι όπου διατέθηκαν τα περισσότερα κονδύλια του κοινωνικού ταμείου. Και είναι σημαντικό για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών. Και επίσης η εδαφική συνεργασία κάνει πολλά ιδίως με την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών στον χώρο της ε, δημογραφικής αλλαγής. Υπάρχει το πρόγραμμα Interreg που λέγεται DART, το οποίο είναι στοχευμένο ακριβώς στη δημογραφική αλλαγή για να φέρει σε επαφή περιφέρειες των ανατολικών ευρωπαϊκών χωρών με δυτικές για να μπορέσουν να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις. Και όταν τα συζητήσαμε αυτά με τους ανθρώπους με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή και τους λάβαμε συνεντεύξεις στη Ρουμανία, είδαμε ότι ήταν πολύ χρήσιμα αυτά τα πράγματα για αυτούς για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στο τοπικό επίπεδο. Βέβαια, δεν υπάρχει μια συνεχτική στρατηγική για τη δημογραφική αλλαγή. Σε ορισμένες λίγες μονοχώρες υπάρχει μια γενικότερη στρατηγική για την ε, αντιμετώπιση δημογραφικής αλλαγής, όπου να βάζει να εργαστούν και να συνεργαστούν όλοι οι ε, σχετικοί φορεί. Και δεν υπάρχει και πλήρη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν τα ταμεία. Δηλαδή κάνουν κάτι χωρίς ωστόσο να στείλουν στα πόδια της μια πραγματική στρατηγική. Υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα, πιθανότατα που μπορούν να γίνουν για τα θέματα αυτά. Επίσης, τα δύο βασικά προβλήματα συχνά διαπιστώνουμε ότι πρόκειται κατακαιρματισμένα μέτρα. Δεν υπάρχει, όπως έλεγα πριν, μια συνολική στρατηγική. Επίσης δε, η βιωσιμότητα των ε, έργων είναι πολύ περιορισμένη, διότι συχνά πρόκειται για πολύ μικρά έργα, project, που όταν πάυσει χρηματοδότηση αυτά αποθνίσκουν. Δεν συνεχίζονται δηλαδή. Όταν κάναμε τα interview για την προγραμματική περίοδο, τότε η προγραμματική περίοδος 2020 βρισκόταν ακόμη στην αρχή τη Προσπαθούσαμε να κατανοήσουμε εμεί εάν η δημογραφική αλλαγή ήταν ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντα στο τοπικό επίπεδο και όσοι, όλοι όσοι τους λάβαμε συνεντεύξεις μας είπαν ότι είναι ένα σημαντικό θέμα και προσπαθήσαμε λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Τα όσα έγιναν τα βλέπετε εδώ. Τα περισσότερα από τα διαφθορτικά ταμεία αφιερώθηκαν στην βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση για ηλικιωμένους, γυναίκες, νέους και μετανάστες. Το δεύτερο ήταν οι κοινωνικές υποδομές, δεύτερος χώρος παρεμβάσεων, δηλαδή σε ό,τι αφορά το ποσό των κονδυλίων που διατέθηκαν για θέματα που έχουν σχέση με τη δημογραφική αλλαγή, επίσης ζητήματα αναζωογόνησης αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου το ίδιο είδαμε λίγες μόνο να πάνε σε πολύ, λίγα μόνο κονδύλια να πάνε σε πολύ περιφερειακές περιοχές κυρίως Φιλανδίας και Σουηδίας που είναι πάρα πολύ απομακρυσμένες. Επίσης, για να προσπαθήσω να ολοκληρώσω έτσι ώστε να προλάβω να σας τα πω όλα μέσα στα 10 λεπτά που με έχετε δώσει, μια στιγμή Λίγα λόγια για το σχέδιο νομοθετικών μέτρων 2014 έως 2020. Το πακέτο αυτών μέτρων δείχνει ότι ακόμα και αν η δημογραφική αλλαγή δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των οριζόντιων στόχων της νέας πολιτικής συνοχής, ωστόσο είναι πολύ περισσότερο στοχευμένη τώρα η πολιτική αυτή από ό,τι ήταν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο μετα... αναφέρεται στο κοινό, στρατηγικό, στο πλαίσιο στρατηγικής. Η αρχή της εδαφικής συνοχής που είναι στη βάση αυτής της νέας πολιτικής συνοχής είναι πολύ σημαντική για να αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές προκλήσεις διότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ειδικέ προκλήσεις των διαφόρων περιοχών διότι βλέπουμε όπως είπα και πριν ότι υπάρχει μεγάλη ετερογένεια μεταξύ των περιφερειών. Ο νέος κανονισμός του Περιφερειακού Ταμείου και του Κοινωνικού Ταμείου στοχεύουν περισσότερο στην ε, βιώσιμη αστική ανάπτυξη με ειδικά καθορισμένη χρηματοδότηση, για ειδικού σκοπούς δηλαδή, καθώς και για ε, περιοχές με πολύ αραιό πληθυσμό, ιδίως για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ίσως που είναι πολύ σημαντική, αλλά ταυτόχρονα και σε μέτρα κοινωνικής συμπερίληψης. 20% του κοινωνικού ταμείου θα πρέπει να πάει σε τέτοια μέτρα κοινωνικής συμπερίληψης. Πάλι εδώ λοιπόν μπορούμε μέσω αυτού να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής. Υπάρχουν και ορισμένα εργαλεία τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό και τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην ε, υιοθέτηση μια κοινή προσεγγίσεως, τοπική ανάπτυξη, ειδικέ ολοκληρωμένες ε, περιφερειακές επενδύσεις μέσα σε ένα συνολικό σχέδιο, γιατί μεταξύ των καλύτερων πρακτικών ήταν και η ικανότητα να ενταχθεί η πολιτική της συνοχής με εθνικές και περιφερειακές πολιτικές και πάλι μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Αγροτικό Ταμείο. Και με αυτή τη συντονισμένη προσέγγιση διαπιστώνουμε ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα και πολύ ισχυρότερα από ότι αν λειτουργήσει ο κάθε από αυτούς τους θεσμούς μόνος. Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω τώρα. Τα διαθωτικά ταμεία και η πολιτική συνοχή είναι από τα πιο βασικά εργαλεία για την στήριξη των περιφερειών για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις αλλαγές, στις δημογραφικές αλλαγές και λόγω κοινωνικής πολιτικής αλλά και διότι η προσέγγιση είναι πολυετής. Δίνει τον χρόνο δηλαδή να γίνουν και διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Όμως η εμπειρία που έχουμε συλλέξει ως τώρα δείχνει ότι δίνεται όλο και μεγαλύτερη προσοχή στα θέματα αυτά, όμως τα μέτρα που λαμβάνονται εξακολουθούν να είναι κατακαιρματισμένα και υπάρχει και πρόβλημα βιωσιμότητας των μέτρων. Για να βελτιώσουμε λοιπόν την αποτελεσματικότητα της ε, περιφερειακής πολιτικής, της συνοχής χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο ευρωπαϊκό επίπεδο στην δημογραφική αλλαγή ένα από τα πιο σημαντικά οριζόντια θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτική της συνοχής με κοινέ αρχές παρέμβασης και στόχους. Δηλαδή οι περιφέρειες θα πρέπει ρητά να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά και είναι απαραίτητο να ενισχυθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ένα, μέσα σε ένα πλαίσιο πολυεπίπεδο διαχείρισης με συμμετοχή των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης, των ταμείων δηλαδή. Και ταυτόχρονα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε κοινοπραξίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Πάλι μεταξύ των βέλτιστων πρακτικών, ορισμένες διαπιστώσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες γιατί είχαν την ικανότητα να ενεργοποιούν και ιδιωτικούς φορείς να παρέμβουν δηλαδή στο επίπεδο της προσπάθειας αντιμετώπισης της δημογραφικής αλλαγής. Επίσης πρέπει να ενισχυθούν νέες προσεγγίσεις που να είναι πιο ενεργές με την έννοια ότι η δημογραφική αλλαγή δεν πρέπει να θεωρηθεί μοναχά ως πρόβλημα αλλά και ως ευκαιρία που θα δώσει λοιπόν την ευκαιρία να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες, να ανοίξουν νέες αγορές, μπορεί να δημιουργήσει κιόλα νέες αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, οι μετανάστες μπορούν να γίνουν και οικονομικοί φορείς και όχι μονάχα απολύπτες της κοινωνικής ενίσχυσης. Έχουν και δεξιότητες, έχουν και ικανότητες που αν αυτές αξιοποιηθούν μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι πρέπει να αναπτύξουμε τη νέα αυτή νοοτροπία σχετικά με τις νέες αυτές αλλαγές και ταυτόχρονα να λάβουμε υπόψη τις νέες οπτικές, τις νέες προσεγγίσεις, ιδίως δε ε, οι τοπικοί θεσμοί πρέπει να αντιληφθούν και να μάθουν πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτά. Και για να αυξηθεί η θεσμική ικανότητα στο περιφερειακό επίπεδο χρειάζεται στήριξη εκ των άνω. Να μάθουν λοιπόν οι θεσμοί αυτοί πώς μπορούν να βελτιώσουν τα πράγματα αυτά. Το ίδιο πρέπει να βελτιωθεί η παρακολούθηση και η υποπτία με συλλογή νέων δεδομένων, και στο περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο για να μπορούμε να αξιολογήσουμε πού ακριβώς εντοπίζονται τα συγκεκριμένα προβλήματα σε κάθε επίπεδο παρέμβασης. Τελευταίες δύο διαφάνειες, το ποιο μπορεί να είναι ο ρόλος των θεσμών της Ένωσης και πιο συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να προσφέρουν και να διασφαλίσουν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων πολιτικών που εφαρμόζονται στο τοπικό επίπεδο να ενισχύσουν τις συνεργασίες, να προωθήσουν και μια συζήτηση βασισμένη σε στοιχεία, γιατί υπάρχει ακόμα πολύ λίγη αξιολόγηση των, ε, της αποτελεσματικότητας των πολιτικών που αντιμετωπίζουν τη μορφική αλλαγή. Και αν δεν υπάρξει αυτό, όλοι συνεχίζουν κάποιες προσεγγίσεις που δεν γνωρίζει κανείς τι αποδίδουν. Άρα χρειάζεται περισσότερη έρευνα και αξιολόγηση των ειδών εκείνων πολιτικής που φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικά. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αναπτυχθούν δεδομένα και δείκτες και να προσφερθεί και στήριξη σε τοπικούς θεσμούς και τοπικούς φορείς έτσι ώστε να είναι πιο προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν τα διάφορα θέματα που προκαλεί η δημογραφική αλλαγή. Τέλος, για το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι εκπροσωπεί τους πολίτες και μπορεί επομένως να δώσει όθηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Επιτροπή Περιφερειών, ώστε τα όργανα αυτά να εγκύψουν περισσότερο στα προβλήματα αυτά πιο έντονα και μπορεί επομένως να ζητήσει από μια χώρα μέλος ή τις χώρες μέλη ή τις περιφέρειες να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στις δημογραφικές προκλήσεις και στις ε, συμβάσεις συνεργασίας, partnership contacts, να ζητήσουν από τις χώρες μέλη να προσφέρουν τεχνική στήριξη και τεχνογνωσία στις περιφερειακές και τοπικές αρχές αλλά και στους τοπικούς φορείς για το πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά. Μπορεί να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από χώρες μέλη να συλλέξουν συγκρίσιμα δημογραφικά δεδομένα, ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να τονώσει την συζήτηση και την συνειδητοποίηση για τα θέματα αυτά. Των διαφορετικών πτυχών, δηλαδή των δημογραφικών προκλήσεων και των τρόπων με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπιστούν. Για παράδειγμα, με την ίδρυση θεματικών σεμιναρίων, άλλων σεμιναρίων και στο ευρωπαϊκό και στο περιφερειακό επίπεδο μπορούν να προκαλέσουν συζήτηση ε, και να ε, εμφυσίσουν ζωή στις συζητήσεις και μεταξύ των ε, πολιτών στην περιφέρεια. Μπορούν και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές να συνεργαστούν με άλλες επιτροπές που ασχολούνται με ε, θέματα δημογραφικής αλλαγής με την ε, Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών, ε, την Επιτροπή Ανάπτυξης και ούτω καθεξής. Και βεβαίως και με την Επιτροπή των Περιφερειών. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και ζητώ συγγνώμη αν θεωρείτε ότι μακρηγόρησα. Δυστυχώς θα πρέπει να ζητήσω από τους επομένους ομιλητές να είναι πολύ πιο σύντομοι. Ο κύριος Άλμπερτ Εστέβε Παλός έχει το λόγο. Hola. Hola. Muy buenas Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμεριστώ μαζί σας την άποψη που έχω για την ευρωπαϊκή δημογραφία και ιδιαίτερα για την προοπτική την οποία παρουσιάζει στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ξεκινήσω χαρακτηρίζοντας δημογραφικά αυτή την περιοχή του νότου της Ευρώπης, παρουσιάζοντας ορισμένα βασικά δεδομένα. Οι χώρες αυτές ε, χαρακτηρίστηκαν και χαρακτηρίζονται ε, σαν χώρες με ιδιαίτερα χαμηλή γονιμότητα. Οι γυναίκες κατά μέσο όρο έχουν κάτω του 1,5 παιδιά η κάθε γυναίκα. Χαρακτηρίζονται επίσης σαν χώρες οι οποίες έχουν ε, αρκετά ιδιαίτερα υψηλή ε, προσδοκία ζωής, 78-79 έτη για τους άνδρες και οι γυναίκες ε, ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν λοιπόν χώρες, βλέπουμε ότι είναι χώρες με χαμηλή γονιμότητα και με υψηλό προσδόκιμο. Και ταυτόχρονα είναι χώρες οι οποίες τα τελευταία 10 χρόνια έχουν δεχθεί και πάρα πολλούς ξένους πολίτες δεν έχω τον χάρτη, αλλά θα μπορούσα να σας δείξω ένα χάρτη ο οποίος δείχνει ότι η Ισπανία και η Ιταλία κυρίως και η Πορτογαλία έχουν ε, δεχθεί πολλούς μετανάστες από το 1998 μέχρι το 2007. Οι χώρες αυτές ε, δυστυχώς χαρακτηρίζονται και από άλλα πράγματα, δυστυχώς επαναλαμβάνω, κάποια επίπεδα ανεργίας πολύ υψηλότερα από τους υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 25% σαν παράδειγμα ανεργία στην ε, Ισπανία. Και ταυτόχρονα οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από ποσοστά ανεργίας των νέων ιδιαίτερα υψηλά. Ιδιαίτερα υψηλά στην Ισπανία το 50% των αγοριών και των κοριτσιών, γύρω στα 25, είναι στην ανεργία. Κάτι το οποίο επίσης μας εκπλήσει είναι ότι οι χώρες αυτές έχουν ένα ποσοστό απασχολουμένων από τις ηλικίες 55 μέχρι 65 ετών που είναι κάτω του 50% και αυτό εκπλήσει. Δηλαδή χώρες οι οποίες έχουν λίγα παιδιά, χώρες που ζουν πολλοί οι πολίτες τους, χώρες που λίγοι δουλεύουν, όπου τα επίπεδα ανεργίας είναι πάρα πολύ υψηλά, τα επίπεδα ανεργίας στους νέους είναι εξαιρετικά υψηλά και τα επίπεδα ανεργίας σε αυτούς που είναι από 55 με 65 έχουν ιδιαίτερα χαμηλά και αυτή επίπεδα απασχολησιμότητας. Τι ακριβώς φαίνεται ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Φαίνεται ότι δεν θα ανακάμψει η γονιμότητα. Έχουμε ήδη όπως είπα χαμηλή γονιμότητα και είχαμε σε περιόδους υψηλής οικονομικής ανάπτυξης. Ε, τώρα με την κρίση δεν θα αυξηθεί. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι υπάρχει ένας, μια αλλαγή στον κύκλο το μεταναστευτικό. Δεχθήκαμε πάρα πολλούς μετανάστες και τώρα βλέπουμε ότι περισσότεροι φεύγουν από τις χώρες αυτές παρά έρχονται. Είναι επίσης πάρα πολύ πιθανό ότι τα επόμενα δέκα χρόνια θα υπάρξει μείωση του πληθυσμού. Είναι επίσης πάρα πολύ πιθανό ότι σε όλες αυτές τις χώρες για τις οποίες μιλάω τώρα τα επόμενα δέκα έτη, στην Ισπανία σαν παράδειγμα το 2017 θα υπάρξουν περισσότεροι θάνατοι από ό,τι γεννήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια αλλαγή δημογραφικού σεναρίου, ουσιαστικά καθοριστική. Στα πλαίσια αυτής της καταστροφικής κατάστασης ε, επιβεβαιώνεται δυστυχώς κάποια γεγονότα, βλέπουμε στον τύπο ότι τίθενται πολλές ερωτήσεις για το μέλλον τι θα γίνει με την κοινωνία μας όταν μειωθεί ο πληθυσμός. Αυτό θα είναι κακό γενικά για τον πληθυσμό. Η δεύτερη ερώτηση που τίθεται είναι τι θα γίνει με τους μεταναστευτικούς κύκλους. Θα αναγκαστούν οι ικανοί προς εργασία να φύγουν από τη χώρα. Και η τρίτη ερώτηση είναι αυτή η οποία ακούγεται πιο πολύ αν θέλετε. Ποιος θα πληρώσει τις συντάξεις αν είμαστε υπερήλικες, δεν υπάρχουν παιδιά και δεν έχουμε και δουλειά, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πληρώνει τις συντάξεις. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε, να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Η πρώτη είναι τι θα συμβεί όταν ένας πληθυσμός συνεχίζει να μειούται. Ε, θα έλεγα ότι δεν συμβαίνει σε μία πρώτη φάση τίποτα το σοβαρό δεν θα πρέπει να μας ενοχλήσει ιδιαίτερα η μείωση του πληθυσμού εμείς θα πρέπει ίσως και να χρειαστεί να εγκαταλείψουμε κάποιες ιδέες οι οποίες μας έχουν καθίσει θα έλεγα τα τελευταία χρόνια όπως το ιδανικό ε, της γονιμότητας. Το θεωρητικό 2,1 παιδιά ανά γυναίκα σαν παράδειγμα. Κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να κρατήσουμε τον πληθυσμό υποτίθεται στο ίδιο επίπεδο. Όχι αυτό είναι ένας μύθος ε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν πεθαίνουν πολλοί, πάλι θα μείνει ε, σταθερός ο πληθυσμός, ακόμα και αν υπάρξουν θάνατοι με τις γεννήσεις, πάνω κάτω πάλι θα διατηρηθεί ο πληθυσμός. Το θέμα είναι ε, σημαντικό να συνδέσουμε τον αριθμό των παιδιών με το προσδόκιμο ζωής των παιδιών αυτών ζώντας περισσότερο τα παιδιά αυτά, αυξανωμένου του προσδόκιμου, με λιγότερα παιδιά, θα διατηρήσουμε προφανώς το ίδιο επίπεδο πληθυσμού. Και αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Νομίζω ότι η Ευρώπη ιστορικά ήταν πρωτοπόρο στην διατήρηση ενός συστήματος αναπαραγωγής που θα χαρακτήριζα πολύ παραγωγικό. 2,1 λοιπόν παιδιά από τις γυναίκες της Ευρωπαίες και διατηρήθηκε το επίπεδο του πληθυσμού όχι μόνο χάρη στη μετανάστευση αλλά και από το ότι υπάρχει μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Είναι απαραίτητο λοιπόν για να διατηρηθεί η κατάσταση αυτή αυτά τα λιγότερα παιδιά τα οποία γεννούνται να είναι πιο παραγωγικά και οικονομικά ένας εργαζόμενος σήμερα στον τριτογενή τομέα να μπορεί να συντηρήσει τέσσερις συντάξεις του πρωτογενού τομέα ε, οι οποίοι έχουν εργαστεί πάνω από 30 χρόνια. Λοιπόν, αν μπορέσουμε εμείς να διασφαλίσουμε ότι κάθε νέα γενιά είναι παραγωγικότερη της προηγούμενης, αυτή η αποκαλυπτική εικόνα της δημογραφικής εξέλιξης είναι λανθασμένη, θα αποδειχθεί λανθασμένη. Δεν νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται εμείς να τονώσουμε με κάποιο τρόπο την ε, γονιμότητα για να έχουμε περισσότερα παιδιά. Να έχουμε περισσότερα παιδιά. Όχι όμως για να έχουμε μια δημογραφική δομή η οποία να πληρώνει τις συντάξεις, αλλά για να δώσουμε τη δυνατότητα στους άνδρες και τις γυναίκες που θέλουν να έχουν παιδιά να το κάνουν και όσα θέλουν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν το ίμιση περίπου αυτών που γεννιούνται σήμερα θα ζήσουν πάνω από 100 χρόνια. Η μισή από αυτούς που γεννιούνται τώρα. Εμείς ταυτόχρονα βλέπουμε ότι τα παιδιά μας τα κάνουμε από τα 25 μέχρι 45 ετών. Αυτό σημαίνει λοιπόν το να είναι κανείς νέος σε μία εποχή, σε μία περίοδο που οι οικονομικές συνθήκες είναι χάλια, σε αυτή την περίπτωση οδηγεί αν θέλετε να μην κάνουν παιδιά και να ζουν με 100 σχεδόν χρόνια από εδώ και πέρα, αλλά χωρίς να αναπαράγονται και χωρίς να αναπαράγονται όχι μόνο διομογραφικά αλλά και κοινωνικά θα έλεγα. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να πείσουμε ότι ο κόσμος που θέλει να κάνει παιδιά μπορεί να τα κάνει παιδιά και όχι λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης να μην το κάνει αυτό. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά την λεγόμενη μακροδημογραφία, αλλά την καθημερινότητά τους, τη ρουτίνα τους, τη ζωή τους. Τώρα, <clears throat> σχετικά με τη μετανάστευση. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα και αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι πράγματι πολλοί Ισπανοί και Ιταλοί το σκέφτονται και βλέπουμε ότι η πλειοψηφία αυτών οι οποίοι φεύγουν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ε, οικονομικές προοπτικές στη χώρα τους, δεν ε, ήταν ικανοποιημένοι οικονομικά και γι' αυτό αναγκάζονται να πάνε σε άλλες χώρες, σε τρίτες χώρες. Δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, μια, ένα μεγάλο ποσοστό ε, αυτοχθόνων που να μετακινείται. Και αυτό δεν θα έχει ιδιαίτερα μεγάλες επιπτώσεις. Είναι σημαντικό επίσης η εμπειρία, η μεταναστευτική την οποία βιώσαμε τα τελευταία χρόνια να μην επηρεάσει την σχέση ανάμεσα στη δημογραφία και την ίδια τη μετανάστευση. Ορισμένοι ειδικοί λένε ότι αυτή τη στιγμή ε, αλλάζει δημογραφικά η Ισπανία ή μπορεί να αλλάξει δημογραφικά η Ισπανία και αυτό θα επιτρέψει να αυξηθεί το ρεύμα των μεταναστών προς την χώρα αυτή. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ακριβώς ε, η όταν υπάρχουν πολλοί Ισπανοί οι Ιταλοί, Ιταλοί Ιταλοί και Ισπανοί Ισπανοί εννοώ, όταν βρίσκουν δουλειά τότε έρχονται πάρα πολλοί μετανάστες. Και έρχονται πολλοί μετανάστες για τον απλούστατο λόγο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις γενιές υπάρχει ευκαιρία και υπάρχει δουλειά για όλους. Αυτό δεν ίσχυε εν πάση περιπτώσει στη δεκαετία του 80. Σαν παράδειγμα. Δεν υπάρχει μια αυτόματη σχέση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στη δημογραφική δομή και την άφηξη των μεταναστών, αλλά μια σχέση οργανική ανάμεσα στην άφηξη των μεταναστών και στην οικονομική κατάσταση. Τώρα να μιλήσουμε τώρα το τι θα γίνει με την γύρανση του πληθυσμού και το ποιος θα πληρώσει τις, α, τις συντάξεις. Κοιτάξτε, απλά έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Είναι καλό νέο αυτό. Έχει αυξηθεί το καλό νέο αυτό λοιπόν κατά τέσσερους μήνες αναμήνα ζωής. Σημαντική αύξηση δηλαδή. Κάθε δέκα χρόνια πάνω κάτω κερδίζουμε δηλαδή δύο χρόνια ζωής. Προσδοκίμου, εν πάση περιπτώσει ζωής. Δηλαδή οι 24 ώρες μας της καθημερινότητας γίνονται 27 ώρες, 30 ώρες σε προσδόκιμα ζωής. Και εδώ οδηγούμεθα στην σχέση, στην ιδέα της αντιμετώπισης της ηλικίας σαν κάτι το ευέλικτο. Η ζωή και η πόλη όπως ζούμε σήμερα δεν θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον. Κάποιος ο οποίος σήμερα είναι 65 ετών δεν είναι κάποιος που θα έχει 65 έτη σε 30 χρόνια. Δεν θα είναι ο ίδιος άνθρωπος, θα είναι διαφορετικός και δεν αισθάνεται ο 65 σήμερα με τον τρόπο που θα αισθάνεται ο 65 μετά από 30 χρόνια. Δεύτερον, το θέμα της αύξησης του προσδόκιμου είναι κάτι το οποίο στην ουσία ε, μας οδηγεί στο να ζήσουμε στον πολίτη μας, ε, στον πλανήτη μας, συγγνώμη, πολύ περισσότερο χρόνο με τους προγόνους μας, με τους πατέρες μας, με τους παππούδες μας, με τους προπάπους μας. Αυτό κοινωνικά προπαλεί πάρα πολλές αλλαγές. Ε, δηλαδή οδηγούμεθα αυτή τη στιγμή σε οικογένειες τεσσάρων γενεών. Δηλαδή παιδιά, πατέρες, παππούδες και προπαππούδες. Βλέπουμε λοιπόν ότι συμπίπτουμε χρονικά Αυτό δεν ίσχυε στο παρελθόν και στο μέλλον θα έχουμε επίσης πολλά περισσότερα παιδιά με προπαπούδες από ό,τι σήμερα. Αυτό δημιουργεί ένα σύστημα κάθε της αρρωγής ανάμεσα στις οικογένειες που οι νέοι με τη σειρά τους θα βοηθούν τους μεγάλους και όταν οι μεγάλοι στην ηλικία έχουν σωρεύσει πλούτη και ικανότητες και δυνατότητες θα βοηθήσουν επίσης τους νεότερους. Δηλαδή δημιουργείται ένα κεφάλαιο και στις ε, μεγάλες ηλικίε και έτσι οι νεότεροι και σε επίπεδο ιδιωτικό, οικογενειακό και σε επίπεδο δημόσιο, μέσα δηλαδή στις δυνατότητες τις οποίες παρουσιάζει η κοινωνία αποκτούν παραγωγικές ικανότητες που με τη σειρά τους θα βοηθήσουν να καλύπτουμε τα έξοδα ε, της, ε, ε, των συντάξεων. Μιλάμε για τον, νόμο της, για τον νότο της Ευρώπης όπου οι σχέσεις οικογενειακές παίζουν πολύ μεγάλη σημασία και θα δημιουργηθούν στο μέλλον ακόμα πιο ισχυρά οικογενειακά συστήματα που θα βοηθήσουν. Λοιπόν, και έτσι ε, αυτό για να γίνει βέβαια θα πρέπει οι τελευταίες γενιές να μπορέσουν να έχουν τις δυνατότητες αυτές. Τώρα για το ποιος θα πληρώσει α, τις συντάξεις, κοιτάξτε. Οι συντάξεις αυτές θα πρέπει πράγματι να προσαρμόζονται στη δημογραφική πραγματικότητα και όχι η δημογραφική πραγματικότητα να προσαρμόζεται στο επίπεδο των συντάξεων. Θα πρέπει να αποφύγουμε να μετράμε το πόσοι εργάζονται και το πόσοι συνταξιοδοτούνται. Αυτή η καταμέτρηση από μόνη της δεν φτάνει. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε το πώς μπορεί ο καθένας συνεισφέρει και πόσο μπορεί να παράγει και να βοηθήσει τη λειτουργία του συστήματος. Θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και τότε δεν θα πρέπει να ανησυχήσουμε για την μείωση του ε, ενεργού πληθυσμού. Έχει όμως πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όπως είδαμε προηγουμένως, να αυξήσουμε τα λεγόμενα επίπεδα απασχολησιμότητας και μάλιστα της λεγόμενης διαγενειακής απασχολησιμότητας. Οι γενιές οι οποίες γεννιούνται σήμερα, οι περισσότερες από αυτές, θα φτάσουν όπως είπα τα 100 χρόνια ζωής και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση το 55% των ανθρώπων αυτών να εργάζονται. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σήμερα και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί με τον τρόπο αυτό. Αν τα αλλάξουμε όλα αυτά, τότε ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε το ποιος θα βοηθήσει ποιον θα αλλάξει. Δεν υπάρχει λοιπόν ουσιαστικά κίνδυνος δημογραφικός, υπάρχει κίνδυνος οικονομικός, θα πρέπει εμείς να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, να αντιστρέψουμε την πορεία, να βελτιώσουμε τις αμοιβέ και το, η Ευρώπη η οποία είναι γνωστή για το παραγωγικό της σύστημα να συνεχίσει να το κάνει με λιγότερα παιδιά ίσως από ό,τι στο παρελθόν αλλά με υψηλότερη παραγωγικότητα διατηρώντας και το επίπεδο της ε, πληθυσμιακής κατάστασης σε κάθε χώρα και την ευημερία της κάθε χώρας. Πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε κάποιες νέες παραμέτρους δημογραφικές. Ζούμε μια νέα μορφή της δημογραφίας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε προβολές ε, στο μέλλον, αλλά να, ε, να μην λαμβάνουμε κάποιες ευέλικτες αλλαγές υπόψη να μην θεωρούμε ότι να μην ξεχνάμε ότι κάποιος ο οποίος σήμερα είναι 70 ετών και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο 70 σήμερα δεν θα είναι η ίδια κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται μετά από πολλά χρόνια. Το θέμα δεν είναι δημογραφικό, το θέμα είναι πολιτιστικό και κυρίως οικονομικό. Θέλουμε λοιπόν οι νέες γενιές οι οποίες ζουν με τις οικογένειάς τους να αποκτήσουν ικανότητες για να μπορέσουν να μπουν στην αγορά εργασία σε καλές θέσεις με αυξημένη παραγωγικότητα. Και ζητάμε να βοηθήσουμε ιδιαίτερα αυτούς που είναι 35-40 χρονών που έχουν δουλειές αλλά των οποίων η κατάστασή τους δεν τους ικανοποιεί και δεν τους οδηγεί να κάνουν παιδιά να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους γιατί όπως είπα μιλάμε για προσδόκιμα ζωής πάρα πολύ υψηλά, κάτι το οποίο θα επηρεάσει ε, στο μέλλον αναγκαστικά ε, την ευημερία όλων. Λοιπόν, ελπίζω να σας μετέφερα, να σας προκάλεσα την προσοχή, μας, να, την προσοχή σας, να σας μετέφερα τις απόψεις μου και δεν πρέπει να ανησυχούμε για τα βιογραφικά, τα δημογραφικά θέματα έτσι όπως παρουσιάζονται, αλλά κυρίως για το οικονομικό κομμάτι. Ευχαριστούμε, ο Λάζ Ράντεμάχερ. Ja, vielen Dank. Ähm, Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Πρόεδρε. Στα γερμανικά. Ευνηδιάζομαι λίγο, εκπλήσωμαι λίγο που βρίσκομαι εδώ, διότι τόσο συχνά δεν συμβαίνει σε επιστήμονα επικοινωνιών να έρθει να μιλήσει για, να προσκληθεί να μιλήσει για ε, δημογραφική συνοχή θα σας σερβίρω λοιπόν κάπως πιο ελαφρά δέσματα. Η μελέτη που με απασχολεί εδώ είναι η στήριξη, ενίσχυση γυναικών που ιδρύουν επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνοδεύσουν τις γυναίκες στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα δομές οι οποίες να μπορέσουν να τις στηρίξουν στα πρώτα βήματα του επιχειρήν. Γνωρίζουμε όλοι ότι η δημογραφική εξέλιξη καθιστά απαραίτητο και οι γυναίκες να εργαστούν επί περισσότερο χρονικό διάστημα και στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μεταξύ αυτών των μέτρων περιλαμβάνεται και η προώθηση συμπεριφορών του επιχειρήν. Μπορεί αυτή η ίδρυση επιχειρήσεων μπορεί να είναι και μια διέξοδος εφόσον δεν λειτουργήσει τόσο πολύ η παραδοσιακή ε, πρόσληψη σε εξαρτημένες ε, εργασίες. Η μελέτη που θα σας υποβαλώ είναι βασισμένη σε μια συνεργασία μετά από πρόταση ενός Συμβουλίου Γυναικών το οποίο συνδέεται με την γερμανική Hypo μεγάλη τράπεζα δηλαδή, που ασχολείται με το πώς αναπτύσσεται η δράση των γυναικών για την ίδρυση επιχειρήσεων και ιδίως εδώ η ιδέα είναι να προσκληθούν γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις επιχειρήσεων να γίνουν οι πνευματικές καθοδηγήτριες, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι, ε, mentor θα έλεγε κανείς για το ανδρικό φύλλο, για να τις καθοδηγήσουν. Αρχικά η χρηματοδότηση ήταν πολύ περιορισμένη. Το ερώτημα λοιπόν ήταν για τη μελέτη πώς θα έλθουμε σε επαφή με τις ε, πολλές γυναίκες. Πρόκειται για μια κοινοπραξία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ε, η οργάνωση αυτή που εκπροσωπείται όμως σε όλα τα ομόσπονδα κρατήδια, ε, βρίσκεται στη Βάδη Βιρτεμβέργη ε, ε, και υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας. Τώρα, η μελέτη πιο συγκεκριμένα. Όλο και περισσότερες γυναίκες ιδρύουν επιχειρήσεις και αυτό μάλιστα αντιβαίνει στην τάση γενικά στη Γερμανία, διότι μειώνεται η ανεργία και παραδοσιακά όταν μειώνεται η ανεργία μειώνεται και η τάση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Όμως είναι σαφές ότι οι γυναίκες ιδρύουν διαφορετικά. Προχωρούν όμως σε αυτό με περισσότερη περίσκεψη, περίσκεψη λιγότερη ανάληψη κινδύνων ε, σε μικρότερα πλαίσια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο επιτυχημένες. Η ιδέα που είχαμε εδώ ήταν να μάθουμε και λίγο περισσότερα πράγματα για την προσωπικότητα των γυναικών που προβαίνουν στην ίδρυση επιχειρήσεων, να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα για το ποια κίνητρα τις ε, παροθούν, που ενδεχομένως ε, σημειώνονται κολλήματα ή φραγμοί. Στην ειδική μελέτη ε, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το mentoring που ανέφερα προηγουμένως. Μεθοδολογικά προχωρήσαμε μαζί με την, με την με τον οργανισμό αυτόν που σας ανέφερα προηγουμένως, που μας έδωσε 8.000 διευθύνσεις και ονόματα ε, των γυναικών εκείνων προς τις οποίες είχε παράσει συμβουλές την τελευταία διετία. Για μετά δεν υπάρχουν δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται συστηματικά. Είναι και δύσκολο λοιπόν κανείς να τα βρει και ε, κυρίως θα είναι πάρα πολύ δαπανηρό κάτι τέτοιο. Επίσης προχωρήσαμε και σε μία υποβολή ερωτήσεων σε mentors, mentors δηλαδή γυναίκες και άντρες και Υπάρχουν και διάφορες παράμετροι, για παράδειγμα, και σφάλματα που ενδεχομένω έχουν γίνει κλπ. Τώρα, για, τα ίδια, για το ίδιο το δείγμα, ερωτήσαμε 424 γυναίκες. Βλέπετε, ούτως ή άλλως, ότι η ηλικία των γυναικών που αναλαμβάνουν την ίδρυση είναι σχετικά υψηλή, δηλαδή 40,5 χρόνια ηλικίας. Ένα πρώτο λοιπόν συμπέρασμα είναι ότι οι γυναίκες προβαίνουν στην ίδρυση επιχειρήσεων ιδίως σε κάπως μεγαλύτερη ηλικία. Οι γυναίκες λοιπόν καταρχήν ιδρύουν αργότερα στην ηλικία, συζητούν, μελετούν, συζητούν με πολλούς τα ε, πιθανά του σχέδια, χρειάζεται δηλαδή και ένα βαθμό ενθάρρυνσης πριν να προχωρήσουν τελικά στην ίδρυση της επιχείρησης. Τώρα, σε ποιους τομείς Ελπίζω ότι φαίνεται η διαφάνεια εδώ. Ο μεγαλύτερος τομέας είναι το κόκκινο, το πορτοκαλί τέλος πάντων, είναι παροχή υπηρεσιών, γενικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών, καθαρισμός κτηρίων, ε, πακέτα υπηρεσιών και βεβαίως σε βιομηχανίες όπως ιατρική, φαρμακευτική κτλ. Στους τομείς αυτούς οι γυναίκες καταρχήν δεν προβαίνουν σε ίδρυση επιχειρήσεων αν και οι ίδιες αυτοχαρακτηρίζονται ως ε, δημιουργικές. Αυτό έχει σχέση και με το μεγάλο αριθμό γυναικών που έχουν μάλλον θεωρητικές ή κοινωνιολογικές ας πούμε σπουδές και προέρχονται λιγότερο από τεχνικούς τομείς ή ε, από τις φυσικές ή θετικές επιστήμες. Άλλοι τομείς που είναι επίσης ισχυροί είναι μεσολάβηση, consulting, διαφήμιση, ε, επικοινωνίες. Επίσης συχνά εκεί ιδρύουν επιχειρήσεις οι γυναίκες. Και, και αυτό έχει σχέση και με προσόντα που θεωρούν οι ίδιες οι γυναίκες ότι διαθέτουν. Και κατά κανόνα αυτές οι ίδιες είναι και ο πυρήνας επιχειρησής τους ή και του προϊόντος τους. Καταρχήν ιδρύουν μόνες τους ή ε, αναδύο. Αναζητούν μία διέξοδο από κάποια πλαίσια που θεωρούν ήταν υπερβολικά δεσμευτικά για αυτές, δηλαδή συνθήκες εξαρτημένης εργασίας, είτε έχουν εγκαταρρύψει τις δουλειές τους διότι δεν μπορούσαν να συμβαδίσουν πλέον με την οικογένεια. Η οικογένεια υπάρχει όμως και γενικά μια έλλειψη ικανοποίησης και επιθυμούν να αναπτύξουν εντονότερα την προσωπικότητά τους. Έχουμε εδώ πάλι μια έντονη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών, να κάνει κανείς σύγκριση με μελέτες του 2012, πάλι για τη Γερμανία, που λένε ότι μέχρι 60% των ανδρών ή του συνολικού δείγματος στη Γερμανία προχωρούν στην είδηση επιχειρήσεων ξεκινώντας από καταστάσεις ανεργίας για τις γυναίκες αυτό είναι διαφορετικό. Εκεί το ποσοστό αυτό των ανέργων γυναικών δηλαδή ανέρχεται μονάχα στο 10% που προχωρούν με τα ίδρυση επιχειρήσεων. Αυτό έχει σχέση όπως είπα και με τους διαφορετικούς στόχους που συνδέονται με την ίδρυση επιχειρήσεων αλλά και με το διαφορετικό προβληματισμό. Οι γυναίκες επίσης είναι πολύ λιγότερο ε, διατεθειμένες να κάνουν συμβασμούς. Πολλοί άνδρες ιδρυτές είναι διατεθειμένοι τα πρώτα χρόνια να κάνουν και σημαντικές παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά την εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, επίσης για τη φροντίδα της οικογένειας, για τις γυναίκες συνήθως δεν συζητείται αυτό. Αυτό για αυτές είναι πάρα πολύ κεντρικό θέμα. Ιδρύουν λοιπόν οι γυναίκες, αλλά μόνο εφόσον έχουν δυνατότητα αυτή. Ρωτήσαμε επίσης την μελέτη μας πώς αισθάνονται μέσα στο υφιστάμενο πλαίσιο ενισχύσεων, πώς δέχονται τις ενισχύσεις για την ίδρυση επιχειρήσεων κλπ. Εκεί οι γυναίκες θεωρούν ότι τις έχει καταλήψει η εξέλιξη. Γυναίκες αναζητούν στοιχεία στα διάφορα προγράμματα ενισχύσεων και των ομόσπονδων και της Ομοσπονδίας και περιφερειακών φορέων Οι γυναίκες δεν λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη σε ό,τι αφορά τις ε, ενισχύσεις που ενδεχομένως δίνονται. Τώρα πάλι σε σύγκριση με άνδρες ιδρυτές νομίζουν οι γυναίκες ότι ο τρόπος συμπεριφοράς των ανδρών ιδρυτών, η μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να παρουσιάζουν το σχέδιό τους απέναντι στους επενδύσεις, ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται απέναντι στους επενδυτές οι άνδρες, αυτό, θεωρεί αυτό θεωρούν μάλλον ότι είναι διαρθρωτικά μειονεκτήματα για τις γυναίκες. Ρωτήσαμε ιδίω εάν οι μέντορες τα ήταν τα πράγματα αυτά διαφορετικά Θέλαμε να γνωρίζουμε δηλαδή αν οι γυναίκε εκεί ίσω είναι ιδιαίτερα επιφρακτικές απέναντι στην ε, δυνατότητα ίδρυση. Οι μέντορε, όχι μόνο επιβεβαίωσαν τι τάσει αυτέ, αλλά μάλιστα θεώρησαν ότι το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο. Η κατάσταση λοιπόν είναι πολύ ε, δυσκολότερη, πολύ χειρότερη από τη, ε, για τις ιδρύτριες δηλαδή από ό,τι οι ίδιες πιστεύουν. Πώς μπορεί να γίνει τώρα επιτυχέστερα αυτό. Πολλές επιχειρήσεις έχουν ε, ασχοληθεί τελευταία να προσφέρουν το mentoring. Είχε ενδιαφέρον για μας να δούμε ότι τα εφιστάμενα προγράμματα είναι σχετικά άγνωστα στο κοινό. Πολλές γυναίκες θα ήθελαν να μπορέσουν να υποφεληθούν, να ζητήσουν δηλαδή και να υποφεληθούν από το mentoring αυτό, δεν γνωρίζουν όμως ποιος το προσφέρει, ποιος είναι ο κατάλληλος συνομιλητής. Ειδικά δε στην Ανατολική Γερμανία είδαμε έναν αριθμό γυναικών που μας είπαν ότι δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη του mentoring. Εκείνες όμως οι οποίες βρίσκονται μέσα σε σχέση mentoring προφανώς επωφελούνται πολύ από αυτό και ιδίως για πράγματα τα οποία χρειάζονται όπως για παράδειγμα υποστήριξη για τα φορολογικά, υποστήριξη για νομικά και οικονομικά θέματα, οι πτυχές της διαδικασίας ίδρυσης και πολύ ουσιώδη πράγματα, αλλά όπως για παράδειγμα τα λογιστικά κτλ. Εκεί δεν βοηθούν μονάχα τα τοπικά επιμελητήρια, αλλά και οι μέντορες αμφωτέρων των φίλων που συνεργάζονται μαζί τους. Ενδιαφέρον ήταν επίσης ότι είδαμε μια σημαντική διαφορά σε ό,τι αφορά την διάθεση προσίδρυσης στη Γερμανία. Το κλίμα, το ιδρυτικό κλίμα το είπαμε εμείς. Οι περιφέρειες εκείνες στη Γερμανία που έχουν ιδιαίτερη οικονομική ισχύ, δηλαδή νότιο-δυτικά. Ε, επίσης η Βαβαρία είναι εκείνες οι οποίε προσφέρουν περισσότερο προσανατολισμό και υποστήριξη στις γυναίκε. Οι ιδρύτριε θεωρούν ότι υποστηρίζονται καλύτερα στον βορρά και στην Ανατολή τη Γερμανία. Αυτό θεωρούν οι γυναίκε. Ίσως επειδή ε, στον νότο τη Γερμανία είναι κάπω πιο παραδοσιακοί οι άνθρωποι σε ό,τι αφορούν την κατανομή των ρόλων των φίλων. Ένα, μια άλλη πτυχή που για μας είχε ενδιαφέρον, όπως είπα από την αρχή, εγώ έχω ασχοληθεί με την επικοινωνία, είμαι επιστήμον της επικοινωνίας και είχε ενδιαφέρον για μένα να δω στην ε, απαρχή αυτή της νέας ε, επικοινωνιακής επανάστασης, να δω πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων λίγο μικρό ρόλο παίζουν τα κοινωνικά δίκτυα για τις ιδρύτριες. Ορισμένες το χρησιμοποιούν αυτό ως marketing platform για να προσφέρουν εκεί προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά όχι περισσότερο, δεν κάνουν άλλη χρήση. Η ιδέα να κάνουν δίκτυα μέσω των ε, κοινωνιακών δικτύων, ε, να αναζητήσουν είτε εταίρους είτε πελάτες, αυτές οι πιθανότητες ήταν πολύ ε, λίγο ανεπτυγμένες στην σκέψη τους. Η δομή των δικτύων δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν τις απασχολεί πολύ. Αυτό θέλουμε εμείς να κοιτάξουμε περισσότερο και να δούμε επίσης κατά πόσο οι γυναίκες εκείνες οι οποίες ίδρυσαν με επιτυχία επιχειρήσεις όντως προχωρούν και στη διαμόρφωση δικτύων. Έρχομαι και στο τέλος της σύντομη αυτής παρουσίασης. Έχω ορισμένα αντίτυπα της μελέτης, θα τα αφήσω στο βάθος της αίθουσας αν σας ενδιαφέρει. Βεβαίως είναι στην γερμανική γλώσσα, αλλά περιλαμβάνει και επισκόπηση στα αγγλικά. Thank you. I, I just wonder whether this is... Σας ευχαριστώ. Δεν λάβαμε την παρουσίασή σας, τις διαφάνειες. Θα μπορούσατε να μας το δώσετε ή να μας το στείλετε με email. θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Και ο συνάδελφος από τη Βαρκελόνη, επίσης καλό θα ήταν αν μπορούσε να μας δώσει την παρουσίασή του, ώστε να υποφελθούν όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ λοιπόν. Ακούσαμε τα αποτελέσματα των μελετών που ζητήσαμε, που ζήτησε το Κοινοβούλιο. Ακούσαμε ε, δύο εμπειρογνώμονες που μας έδωσαν συμπληρωματικά στοιχεία ως προς τα πορίσματα των μελετών. Θα ήθελα να αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση. Ε, Λάμπεχτ, Φανίστερη. Α, η Κίστεν. Οι κυρίες προηγούνται. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είχα την ευχαρίστηση και την τιμή να συντάξω έκθεση πρωτοβουλίας για διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές για τη δημογραφική αλλαγή. Και πολλά από τα όσα άκουσα σήμερα τα περιλάβαμε εκεί και όλα πήγαν σωστά. Και αυτά που είπατε σωστά είναι. Μία από τις δηλώσεις που ήταν πολύ σημαντικές πάντοτε για μας είναι ότι η δημογραφία, η δημογραφική εξέλιξη δεν πρέπει να κριθεί μοναχά ως κίνδυνος αλλά και ως ευκαιρία. Γνωρίζουμε ότι κάθε δεύτερο κοριτσάκι που γεννιέται σήμερα θα φτάσει τα 100 χρόνια. Υπέροχο! Μακάρι και εγώ να φτάσω την ηλικία αυτή, αλλά ή δυνατόν βέβαια σε καλή υγεία. Βέβαια για να γίνει αυτό χρειάζονται και ορισμένα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα και ασχοληθήκαμε στην έκθεσή μας με αυτό και κάτι που μας ικανοποιεί πολύ είναι και στις τελικές διαπραγματεύσεις για την πολιτική συνοχή αλλά και διαδοτική πολιτική είναι ότι αυτό απηχήθηκε μέσα, βρήκε δηλαδή απήχηση. Ενώ στην προηγούμενη περίοδο δεν έπαιζε ρόλο, τώρα αρχίζει και παίζει ρόλο. Και πολλές περιφέρειες το λαμβάνουν υπόψη. Η ίδια προέρχομαι από περιφέρεια γερμανική δηλαδή που είναι αρκετά ευπορή την Βαβαρία δηλαδή αλλά και στη Βαβαρία υπάρχουν περιοχές όπου υπάρχουν ε, βαθιές αλλαγές και όπου ο κόσμος σηκώνεται και φεύγει διότι δεν υπάρχουν ε, θέσεις απασχόλησης, διότι δεν υπάρχουν θέσεις εκπαίδευσης, επαγγελματικής δηλαδή. Και επομένως συγκεντρώνεται ο κόσμος σε αστικά κέντρα και οι άλλοι μένουν μπουκάλες όπως λέμε στα ελληνικά. Υπάρχει λοιπόν το πρόγραμμα αυτό και η βαβαρική κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη, λέει ότι δεν είναι δυνατόν ορισμένες, σε ορισμένες ε, περιφέρειες να υπάρξει πλήρης αφέμαξη και αλλού να υπάρξει τέτοια ε, συγκέντρωση πληθυσμού. Δεν μπορούμε να φέρουμε όλο τον κόσμο στις ε, πόλεις, διότι τότε θα έχουμε πρόβλημα στέγης. Θα χρειαστεί λοιπόν και εκεί να υπάρξει μια διαμόρφωση της ε, ε, δομής των διαθώσεων των πόλεων. Επαναλαμβάνω ότι νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε, συνεχίσουμε να συζητούμε και ταυτόχρονα να συζητούμε με τις περιφέρειες. Λίγα λόγια τώρα για τον αριθμό των γεννήσεων. Μιλήσατε πριν για τον νότο της Ευρώπης. Υπάρχουν όμως και άλλα παραδείγματα στην Ευρώπη που ίσως να μην είναι χώρες που ε, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω όμως την Νορβηγία. Γνωρίζω ότι στην Νορβηγία υπήρξε αύξηση των γεννήσεων. Όμως αυτό έγινε διότι δεν υπήρχε πρόβλημα για τις γυναίκες να συνδυάσουν την επαγγελματική με την οικογενική ζωή. Εκεί λοιπόν από κρατικής πλευράς έγιναν πολλά πράγματα για τη φροντίδα του παιδιού, για την προσφορά σχολικής εκπαίδευσης, για μέτρα υποδομών, έτσι ώστε οι γυναίκες να μπορούν να συνδυάσουν τα δύο. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικά και πρέπει να κινηθούν εκ παραλλήλου. Για να μην μακρηγορήσω λοιπόν, να σας πω μονάχα ένα πράγμα ακόμη για τις γυναίκες ιδρύτριες. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 είχαμε και το πρώτο μεγάλο κύμα ιδρύσεων που πολλές προσπάθησαν να ανεξαρτητοποιηθούν, αλλά λόγω ανάγκης. Πολλές έπεσαν ωστόσο άσχημα, προσγειώθηκαν ανώμαλα. Το μοντέλο των ιδρυτριών λοιπόν ή της ιδρύτριας, μπορεί σε επιμέρους περιπτώσεις να είναι πολύ θετικό. Όμως σίγουρα δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δηλαδή πρέπει να διαμορφώσουμε έτσι την επαγγελματική ζωή ώστε άνδρες και γυναίκες σε οποιοδήποτε φύλου και οποιοδήποτε χρώματος επιδερμίδος να μπορούν να έχουν τις ίσες ευκαιρίες στην ε, πρόσβαση στην εργασία. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, στο τέλος ε, μιας χρονιάς να βλέπουμε τα πορίσματα μελετών που παρουσιάζουν τέτοιο ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία. Εξετάστηκαν οι δημογραφικές τάσεις, αυτό είναι στα μεγάλη πρόκληση, κυρίως για τις ε, συντάξεις, για τη χρηματοδότηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, για τη γύρανση του πληθυσμού, για το ρόλο που πρέπει να αναλάβουν πλέον τα, τα κράτη Ακούσαμε λοιπόν κάποιες παρεμβάσεις από ανθρώπους που πραγματεύτηκαν ε, το ζήτημα των αλλαγών και πώς συνδέεται αυτό με τις νέες πολιτικές. Ε, μου φάνηκαν όλα αυτά και πολύ ενδιαφέροντα και πολύ χρήσιμα. Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα. Ε, μιλήσατε για τον ευθύνοντα πληθυσμό και Ε, συχνά συζητείται αυτό το ζήτημα ε, στην Επιτροπή μας. Ε, επίσης το συνδέουμε με το ζήτημα της μείωσης του εισοδήματος κατά κεφαλή. Όταν μιλάμε για τις δημογραφικές αλλαγές, ταυτόχρονα μιλάμε και για το δυναμισμό των επιμέρους περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον επιμερισμό των πόρων που διαθέτουμε. Πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει κατά τον επιμερισμό των ε, κονδυλίων ε, που διατίθενται στις ε, περιοχές να λαμβάνεται υπόψη η μείωση του πληθυσμού. Έχετε συνυπολογίσει, συνεκτιμήσει όλους αυτούς τους παράγοντες και ποια λύση διαβλέπετε ποιες επιπτώσεις θα έχει η μείωση του πληθυσμού στην επόμενη προγραμματική περίοδο για την πολιτική συνοχή, παραδείγματο χάρη. Τώρα, δεύτερη ερώτηση. Ε, υπάρχουν πολλά νέα προγράμματα για την τεχνολογία της ε, πληροφορίας, ε, της επικοινωνίας. υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που δεν ε, έχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες. Έχουμε νέες δυνατότητες χάρη στους δορυφόρους πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό αλλά για το σύνολο του πληθυσμού διότι μην ξεχνάμε ότι πέρα από τις ωφέλειες που μπορεί αυτό να έχει για τους πολίτες μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και για τις επιχειρήσεις, για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, για την παροχή νέων υπηρεσιών, για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, την τόνωση ε, της απασχόλησης σε μειονεκτούσες περιοχές. Ε, δυστυχώς ε, θα χρειαστεί να αποχωρήσω ευθύ αμέσω, ε, διότι πρέπει να συναντήσω κάποιον. Θα ακούσω όμω, επειδή αναμεταδίδει τη συνεδρίαση, τη απαντήσεως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. και ε, πολύ με ενδιαφέρει ιδίω η δράση αυτού του Ολλανδικού ε, Ινστιτούτου. Δεν ήξερα καν ε, ότι υπάρχει αυτό το Ινστιτούτο και ότι ερευνά τα δημογραφικά ζητήματα. Ε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντοτε να τονίζουμε τις συνέργειες που υπάρχουν ανάμεσα στα εθνικά ερευνητικά ιδρύματα γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε πληροφορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Βίκτορα, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθυνθώ στους διακεκριμένους προσκεκλημένους μας ε, και οι τρεις ε, ομιλητές έκαναν πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις που κάλυψαν τρία, το θέμα σε τρία επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, αποδεικνύεται ότι η δημογραφική κατάσταση της Ευρώπης των 28 κρατών είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και ότι οι προκλήσεις ε, στις οποίες καλούνται οι περιοχές ε, να αντεπεξέλθουν διαφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό εάν ε, συγκρίνουμε την Βαβαρία ή την Σουηδία αφενός και αφετέρου νότιες χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία ή η Ελλάδα διακρίνουμε τεράστιες διαφορές. Δεν είμαι κοινωνιολόγος αλλά μπορώ να σας μιλήσω για τη Ρουμανία, να σας δώσω κάποια στοιχεία τα οποία δεν αναφέρθηκαν, τα οποία όμως είναι χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά ως προς αυτές τις μεγάλες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να προσδιορίσουμε ε, το είδος της κοινωνίας, ε, το κοινωνικού μοντέλου που επιθυμούμε για το μέλλον και το είδος της ανάπτυξης που επιθυμούμε. Καταρχάς, ας αρχίσουμε ε, με τις επιπτώσεις της κρίσης που όξιναν αρνητικές δημογραφικές τάσεις που είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Ε, Στι νότιε χώρε δε ε, μπορεί να αποδοθεί η μείωση του πληθυσμού σε αυξημένε μεταναστευτικέ ε, τάσει των πολιτών, διότι οι πολίτε των νοτίων χωρών πηγαίνουν, μετικούν σε χώρε όπου μπορούν να έχουν μια καλύτερη δουλειά και υπάρχει το γνωστό φαινόμενο που ονομάζεται διαρροή εγκεφάλων, brain drain Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η πολιτική ελίτ αυτών των χωρών ε, πρέπει να υπομειστεί την ε, ευθύνη της ε, διότι στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας, στον επιχειρηματικό κόσμο παρατηρείται η ίδια διαρροή. Αυτό καθ' αυτό το φαινόμενο δεν είναι επικίνδυνο, όμως έχει ιδιαίτερα επικίνδυνες δημογραφικές επιπτώσεις. Ε, τι εννοώ. Ε, εάν συρρυκνωθεί η οικονομία, στο μέλλον ε, θα καταστεί ακόμη δυσχερέστερη εξέβρεση εργασίας, παραδείγματος χάρη, ε, η, ε, η φθήνουσα ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας ε, συνεπάγεται και χαμηλότερο προσδόκιμο. Έχουμε με, στην Ρουμανία τα τελευταία 40 χρόνια τα υψηλότερα ποσοστά εθνισιμότητας λόγω χαμηλών υπηρεσιών υγείας. αν στραφώ τώρα στο θέμα της ανεργίας των νέων, συνειδητοποιούμε ότι οι ελπίδες και η εμπιστοσύνη των γυναικών είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο. Δεν μιλάμε μόνο για την Ισπανία, για την Πορτογαλία, για την Ελλάδα. Αυτό ισχύει και για τη Ρουμανία. Η αυξημένη ανεργία στους νέους ε, έχει ως αποτέλεσμα να μην επιθυμούν οι νέοι να δημιουργήσουν οικογένεια παραδείγματος χάρη. Όλοι γνωρίζουν πόσο κοστίζει το να έχεις οικογένεια. Εάν λοιπόν είσαι άνεργος, ε, σίγουρα διοχετεύεις ε, την ενέργειά σου στην εξέβρεση ε, μιας θέσης εργασίας και όχι στην ίδρυση μιας οικογένειας, κατά προτεραιότητα τουλάχιστον. Απομακρύνονται οι λοιπόν από την ιδέα της ίδρυσης της οικογένειας και προκύπτουν τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων φυσικά. Μειώνεται λοιπόν ο αριθμός των γεννήσεων και ε, απομακρύνεται ακόμη περισσότερο ο απότερος στόχος ε, που είναι η αποκατάσταση των προηγούμενων δημογραφικών τάσεων. Η κατάσταση επιδεινώνεται στην Ήπεθρο, στη Ρουμανία. Αυτή τη στιγμή, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, στην Ήπεθρο οι νέοι ε, έχουν λιγοστές δυνατότητες να ε, φοιτήσουν σε πανεπιστήμια και άρα να έχουν πρόσβαση σε καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Έχουμε επιστρέψει στην κατάσταση δεκαετίας του 30 κάτω από 4% του πληθυσμού των νέων στην Ήπεθρο φυτά στο Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή στη Ρουμανία. Η έλλειψη τέτοιας προοπτικής ε, που έχει φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα πλέον, ε, συνεπάγεται επίσης σοβαρότατη απώλεια ανθρώπινων πόρων και ε, αυξάνεται ο αριθμό των ανθρώπων που δεν διαθέτουν δεξιότητε και άρα μπορούν να στραφούν σε ταπεινωτικέ εισαγωγικά ε, θέσει εργασία ε, που απαιτούν λίγε δεξιότητε και άρα εξωθούνται στην περιφέρεια τη κοινωνία ε, με όλες τις παράπλευρες απώλειες που αυτό συνεπάγεται. Ε, φυσικά αυτό μπορεί να αποδοθεί και στην πολιτική λιτότητα, όπως ανέφερε ο Ισπανός ομιλητής. Ε, η λιτότητα έχει ένα τριπλό στόχο. Πρώτα απ' όλα, μάλλον έχει τρεις επιπτώσεις. Σοβαρές περικοπές στην δημόσια διοίκηση, στον τομέα της υγείας και στον τομέα της εκπαίδευσης. όμως ε, ε, οι δημογραφικές επιπτώσεις ε, αυτής της πολιτικής λιτότητας είναι πάρα πολύ καταστροφικές διότι αλλοιώνεται όχι μόνο η δημογραφική δομή αλλά και το κοινωνικό μοντέλο αυτών των χωρών και ξαναλέω επιστρέφουμε στις αρχές του 20ου αιώνα και όχι στις αρχές του 21ου αιώνα στην εποχή της πληροφορίας και της κοινωνίας της επικοινωνίας και της πληροφορία. Ίσως ε, θα μπορούσαν να ανατραπούν αυτές ε, οι τάσεις ε, με μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής, αλλά σίγουρα κάθε κράτος θα πρέπει να διαθέτει και ίδιους πόρους. Σε κάθε περίπτωση χρειάζονται νέες επενδύσεις σε χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία στα νέα σε εισαγωγικά κράτη-μέλη υπάρχουν στον τομέα της ε, πληροφορικής. Λιγοστοί άνθρωποι με τις απαιτούμενες ε, δεξιότητες ε, είναι ευμετάβλητη η αγορά εργασίας και τελικά δέχονται οποιαδήποτε θέση εργασίας και δεν ε, τελειοποιούν τις δεξιότητές τους. Ε, παραδείγματος χάρη σε μια εταιρεία όπως η Mercedes επενδύει στην Ρουμανία επειδή είναι χαμηλότερες οι αμοιβέ. Εμείς όμως δεν διαθέτουμε πλέον μηχανικούς ή ε, μηχανολόγους διότι έχουν αποχωρήσει και είμαστε καταδικασμένοι στην υπανάπτυξη για το μέλλον. Αυτή είναι μια αλήθεια που δυστυχώς δεν παραδέχονται οι πολιτικοί ε, και αυτό οφείλεται στην έλλειψη, στην ουσιαστική έλλειψη μεταναστευτικής πολιτικής ε, της Ευρώπης. Ενώ είναι αντιμέτωπη με ένα πραγματικό πρόβλημα μετανάστευσης η Ευρώπη. Μπορούμε να παίζουμε και να μαγειρεύουμε τα στατιστικά στοιχεία για όσο χρόνο θέλουμε και μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα στατιστικά στοιχεία ε, για να υποστηρίζουμε τις θεωρίες μας και τους στόχους που εμείς θέτουμε. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Χρειάζομαστε μια ευρωπαϊκή απάντηση για αυτό το πρόβλημα. Ε, είναι γυράσκον ο έχουμε πρόβλημα ενεργού πληθυσμού, είναι ανεπαρκής και δεν μπορεί να καλύψει τις ε, κενές θέσεις. Ε, το δυτικό οικονομικό μοντέλο έχουμε μεγάλο αριθμό μεταναστών από τρίτες χώρες ή ε, ε, μετανάστες που πλέον έχουν ε, πολιτογραφηθεί, είναι νέοι, αν θέλετε, υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θεωρούν αυτούς ως μετανάστες παρόλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση ε, όμως ε, είναι ε, αναμφισβήτητο το ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε διότι ένα μεγάλο κομμάτι του ενεργού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρωτού σημειωθούν όλα αυτά τα μαζικά μεταναστευτικά ρεύματα δεν, θέλει, δεν ήθελε να καλύψει τις κενές θέσεις. Αν εξετάσουμε την ιστορία της ανθρωπότητας μπορούμε να αντλήσουμε διάφορα διδάγματα για αυτά. Πάντως οι δημογραφικές τάσεις σίγουρα μπορεί να αποτελέσουν ένα μεγάλο μεγάλο κόλλημα ε, στην ε, αναπτυξιακή πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα έχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Κίνα, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή ε, μετασχηματίζει το μοντέλο της. Η Κίνα Χρειάζεται ένα συνταξιοδοτικό σύστημα για 800 εκατομμύρια ανθρώπους αυτή τη στιγμή και αναθεωρεί το σύστημα όπως θα έπρεπε να κάνουμε και εμείς ακριβώς τώρα, διότι ε, εάν δεν είμαστε ειλικρινεί, θα βρούμε και ψευδείς απαντήσεις στα προβλήματα που έχουμε. Συγγνώμη που ακριβώ. Ευχαριστώ η Μαρία. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ακτινογραφία την οποία μας παρουσιάσατε και το χάρτη των ευρωπαϊκών πληθυσμών και ιδιαίτερα τον χάρτη των πληθυσμών στις χώρες του Νότου και ιδιαίτερα στην δική μου χώρα, δηλαδή την Ισπανία. Συμμερίζομαι, θέλω να συμμεριστώ την αισιοδοξία σας πέρα από τα ε, ε, ερωτηματικά τα οποία τίθενται σήμερα. Το θέμα είναι τι θα γίνει στο μέλλον και ποια θα είναι η επίπτωση της κρίσης. Ε, γνωρίζω πολύ καλά το τι γίνεται και πόσο μένουν ακριβώς ε, στους, ε, στις οικογένειές τους, συνδέονται όλα αυτά τα προβλήματα με την κατάσταση των νέων. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, σίγουρη σε σχέση με αυτά τα οποία είπατε. Ε, μας έδωσε πρόσφατα η στατιστική υπηρεσία την ακτινογραφία των μεγάλων ισπανικών πόλεων όπου συγκεντρώνεται ο πληθυσμός και σε σχέση με την ε, εδαφική συνοχή και την παρέμβαση του ΦΕΝΤΕΡ και των υπολείπων ευρωπαϊκών ταμείων. Βλέπουμε ότι 1,7 των ε, κατοίκων είναι άνω των 65 ετών. Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς μένουν μόνοι. 1,2 Και τελικά οι στατιστικές υπηρεσίε λένε ότι αυτή τη στιγμή ε, στα τέσσερα άτομα που συνήθως ε, αποτελούσαν ε, την ευρωπαϊκή οικογένεια, την ισπανική οικογένεια, τώρα είναι δύο συνήθως ο πιο συνηθισμένος τύπος της οικογένειας και το 65% των οικογενειών δεν έχει εν πάση περιπτώσει παιδιά στην παρούσα φάση. Αυτές είναι οι επιπτώσεις της κρίσης. Και γι' αυτό θα ήθελα να μάθω εγώ σαν πολιτικός τι προβλέψεις έχουμε, γιατί οι αλλαγές οι οποίες προκλήθηκαν μέχρι τώρα, μέχρι τα τελευταία χρόνια, και όχι μόνο μέχρι το 2008 αλλά μέχρι σήμερα πώς θα αλλάξουν την κατάσταση αυτή της πόλης. Ξέρουμε ότι γυράσκει η Ευρώπη αλλά γνωρίζουμε ότι ο Νότος γυράσκει ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ Μαρία Γεν Νίλσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ σε πολιτικό επίπεδο ήμουνα υπεύθυνο για αυτά τα προγράμματα ε, στην ε, Βόρεια Σουηδία για 20 χρόνια Ενεπλάκιν, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό ε, σε αυτή τη διαδικασία και είδα ποιες είναι οι προκλήσεις για τα κέντρα που διαχειρίζονται τα προγράμματα. Όταν εκπονήθηκαν οι στρατηγικές ε, διαπιστώσαμε ότι ε, τα προγράμματα αυτά δεν συνδέονταν απαραίτητα με τις προκλήσεις που είχαμε εμείς διαπιστώσει σε τοπικά και, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Όμως η κατάσταση αλλάζει ραγδαία. Τα τελευταία 25 χρόνια, παραδείγματο χάρη, έχει μειωθεί πολύ σημαντικά ο πληθυσμός στη Βόρεια και Μέση Σουηδία. Δηλαδή πριν από 100 χρόνια ζούσαν οι άνθρωποι στα δάση. Είναι φυσιολογικό, έχουμε πάρα πολλά δάση εμείς στη Σουηδία. Ε, και ε, έχει αλλάξει η βιομηχανική κατάσταση, δεν ε, δουλεύουν οι άνθρωποι τις ίδιες μηχανές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ευθύνει ο πληθυσμό σε πολλές περιοχές της Σουηδίας. Τα τελευταία 25 χρόνια σημειώθηκαν λοιπόν πάρα πολλές αλλαγές. Στην Βόρεια Σουηδία, παραδείγματος χάρη, έχει η ε, εξορρυκτική βιομηχανία ε, ε, γνωρίζει μεγάλη άνθηση και αυτό τράβηξε πάρα πολλούς ανθρώπους, όμως ήταν fly in, fly out αυτές οι θέσεις εργασίας. Δηλαδή εργάζονταν για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι στα ορυχεία. Ε, στη συνέχεια, ε, ως προς την έρευνα, την ανώτατη εκπαίδευση, υπάρχουν κάποια περιφερειακά κέντρα ε, σε μεγάλες πόλεις, πανεπιστημιακά κέντρα που τραβούν πολλούς φοιτητές. Δεν είναι μεγάλες οι πόλεις, αλλά είναι μεγάλες για την Σουηδία. Αυτό είναι ένα θέλγητρο για τους νέους. Στη συνέχεια ε, υπάρχει μια ιδιαίτερα ε, έντονη μεταναστευτική τάση προς την ε, Σουηδία. Σε μια κρίση όπως παραδείγματος χάρη αυτή της Συρίας υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που χρειάζονται μια νέα πατρίδα και ανοίγει τις αγκάλες της η Σουηδία και τους υποδέχεται. Για μας είναι στρατηγική σημασία στο ζήτημα της μετανάστευσης για αύξηση του πληθυσμού αντικατάστασης του γεράσκοντος πληθυσμού μακροχρόνια. Αυτές είναι οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να σας θέσω την τελευταία ερώτηση. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο στην Ευρώπη οι νέοι ε, σε κάποιες ε, κοινωνίες ψάχνουν μια δουλειά η οποία ουσιαστικά δεν ε, ε, υπάρχει όμως, ενώ σε άλλες κοινωνίες άλλοι θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους δουλειά, θέλουν να είναι αυτοαποσχολούμενοι, θέλουν να φτιάξουν νέες επιχειρήσεις, startups, ε, κυρίως στην Ισπανία βλέπουμε μεγάλη υψηλή ανεργία των νέων. Ψάχνουν δουλειές που δεν υπάρχουν. Ε, μας μιλήσατε για τις οικογένειες τριών γενεών. Το παράδοξο όμως είναι ότι στην Ισπανία οι παππούδες ε, βοηθούν ε, οικονομικά τους νέους που έχασαν τη δουλειά τους ή που δεν είναι άνεργοι ενώ ε, το φυσιολογικό θα ήταν οι νέοι να βοηθούν τους πιο ηλικιωμένους. Είναι νέο αυτό το δεδομένο. Πώς να το αντιμετωπίσει κανείς. Είναι τόσο θετική αυτή η τάση όπως την παρουσιάζεται ή ενδεχομένως να προκύψουν προβλήματα λόγω αυτής. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στους τρεις ομιλητές με όποια σειρά θέλετε, δεν έχουμε πρόβλημα για να κάνετε σχόλια ή να απαντήσετε στις ερωτήσεις που θεωρείτε ότι μπορείτε να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλιά σας. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που ανέκυψαν και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτον, γονιμότητα, ποσοστά γεννήσεων ε, και υποστηρικτικές πολιτικές για την αύξηση του αριθμού γεννήσεων. Μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλουμε περισσότερα παιδιά ή όχι, αλλά τέλος πάντων απόφαση των ανθρώπων είναι. Πρέπει να μπορούν να διαλέγουν πόσα παιδιά θέλουν. Εάν ε, κάνουμε μια συγκριτική μελέτη των ε, εθνικών πολιτικών, στη σελίδα 36 έχετε μια ε, γραφική παράσταση όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι στις βόρειες χώρες και κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες και κυρίως στη Γαλλία είναι υψηλότατα τα ποσοστά γεννήσεων γιατί εκεί υπάρχουν σχετικές πολιτικές που υποστηρίζουν τη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν χωρά συζήτηση. Εάν θέλουμε να αυξηθεί η συμμετοχή ε, των γυναικών στην αγορά εργασίας αλλά και να γεννούν περισσότερα παιδιά πρέπει να στραφούν προς αυτές τις πολιτικές. Δεύτερο θέμα, ε, τεχνολογική καινοτομία. Ε, η τεχνολογία τη σήμερα ημέρα ε, υποστηρίζει νέου τρόπου παροχή υπηρεσιών, ακόμη και σε εξόχω απόκεντρε περιοχέ, ε, υπηρεσίε προ του ηλικιωμένου, ε, προ άτομα με εμποδιζόμενα, με ειδικέ ανάγκε. Μπορούμε να επενδύσουμε ε, ηλεκτρονική ε, εκπαίδευση, ηλεκτρονική διοίκηση. Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτά. Υπάρχουν νέα προϊόντα και νέε υπηρεσίε, νέε αγορέ ε, που μπορούν να αναπτυχθούν, διότι οι ηλικιωμένοι είναι καταναλωτέ επίση και στον τουρισμό. Παραδείγματο χάρη υπάρχουν νέοι τρόποι Μπορούμε να προωθήσουμε προϊόντα για ηλικιωμένου, για εμποδιζόμενου κτλ. Νέε ευκαιρίε λοιπόν παρουσιάζονται. Νέα έρευνα δε για αυτές τις νέες δυνατότητες ε, μπορεί να ε, διεξαχθεί ε, και να τονωθούν οι ανταλλαγές ανάμεσα στα ερευνητικά ιδρύματα και ε, τα ε, ιδρύματα που διαχειρίζονται τα τεκμήρια, τις αποδείξεις, τα στατιστικά στοιχεία που βασίζονται στην πραγματικότητα. Διότι αν δεν υπάρχει αυτή η ανταλλαγή, εκπονεί ο καθένα την πολιτική του, δεν συνεννοείται κανεί με κανέναν, δεν υπάρχει συντονισμό και ε, δεν είναι καλά τα αποτελέσματα. Τρίτον, τα αποτελέσματα της κρίσης. Αυτή η κρίση ήταν η χειρότερη από τη δεκαετία του 30 και δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι η απόλυξή της. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι συγκυριακά μόνο τα αποτελέσματα, ε, αλλά και διαρθρωτικά αρνητικά αποτελέσματα, χαμηλότερος αριθμός γεννήσεων, χαμηλότερο προσδόκιμο επιδείνωση των συνθήκων διαβίωσης. Ας δούμε προς τα πού οδεύει η κοινωνία, αν ε, φτωχαίνουν ε, Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Ε, η μετανάστευση τώρα, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, Υπάρχει το εξή πρόβλημα. Ε, νέοι, νέε με υψηλέ δεξιότητε αποχωρούν από αυτέ τι χώρε, άρα απουσιάζει το εργατικό δυναμικό με ε, υψηλέ δεξιότητε. Σε χώρες όπως ε, στην περίπτωση της Λιθουανίας που σας παρουσιάζουμε στη μελέτη, ε, σχεδιάστηκε μια πολιτική για να προσελκύσουμε νέους με υψηλές δεξιότητες για να επιστρέψουν στην Λιθουανία, να επιστρέψουν μαζί με τις δεξιότητές τους για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Υπάρχουν και σε αυτόν πολιτικές λοιπόν, που έχουν σχεδιαστεί. Αυτοαπασχόληση για τους νέους και τις νέες το πρόβλημα, ε, μάλλον αυτό μπορεί να αποτελέσει λύση, λύση, τέλος μια διέξοδο, αλλά δεν υπάρχει επιχειρηματικό δίκτυο, δεν υπάρχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ε, οι νέοι και οι νέες ε, και κυρίως οι νέες αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερες δυσκολίες ε, για να ιδρύσουν τη νέα τους επιχείρηση, τη δική του επιχείρηση και αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα ποτέ δεν θα έχουν ισότιμες ευκαιρίες οι νέες σε σχέση με τους νέους για να ε, ε, ιδρύσουν δική τους επιχείρηση. Το άλλο πρόβλημα είναι οι ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι τους. Είναι διωγγούμενο το πρόβλημα, αληθεύει ότι ζούμε περισσότερα χρόνια. Επίσης αληθεύει όμως ότι αυξάνεται ο αριθμός ανθρώπων πάνω από 85 χρονών ε, κλινήρει συνήθως και τους φροντίζουν συνήθως γυναίκες. Τι θα κάνουμε. Κάπως πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, διότι είναι μια πραγματικότητα που συνδέεται ε, με τις δημογραφικές αλλαγές. Υπάρχουν ε, οικονομικές προκλήσεις, αλλά το θέμα είναι πως Άρδιν πρέπει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την οικονομική ανάπτυξη της ε, ε, πολιτικές απασχόλησης, εργάζονται περισσότερα χρόνια οι άνθρωποι, οι γυναίκες δεν μένουν στο σπίτι πλέον εργάζονται, χρειαζόμαστε περίθαλψη για τους ε, ηλικιωμένους, ε, χρήση της τεχνολογίας, διαφορετική χρήση των νέων τεχνολογιών για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Ποιος θέλει τώρα να μιλήσει, παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομα. Σχετικά με την έννοια της γονιμότητας. Είναι προφανές ότι είναι απαραίτητες όλες οι πολιτικές που υπάρχουν και που μπορούμε να φανταστήσουμε για να βοηθήσουμε τη γονιμότητα των γυναικών και να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε και τα θέματα του συνδυασμού σαν παράδειγμα της οικογενειακής ζωής με την επαγγελματική κτλ αλλά να μην περιμένουμε παρακαλώ θαύματα από εδώ και πέρα. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δεν έχουν παιδιά πολύ συχνά για τέσσερις χοντρικά λόγους. Καταρχάς υπάρχουν, παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι μάλλον οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν παιδιά. Έχει υπάρξει αν θέλετε μια αλλαγή αξιών ε, θεωρούν ότι τα παιδιά είναι μια δέσμευση σε βάση περιπτώσει. Κάποιοι δεν επιλέγουν τον γάμο αλλά κάποιες πιο ελαστικές μορφές συμβίωσης και θεωρούν ότι η ζωή είναι ωραία και ότι δεν χρειάζεται να δεσμεύονται ε, σε έναν κόσμο με παιδιά. Αυτή είναι μια κατηγορία, ένας λόγος. Υπάρχει άλλη μια κατηγορία που θέλει ε, να έχει παιδιά αλλά δεν έχει πώς να το κάνει. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι δεν συμβιώνουν. Θα πρέπει όπως είπαμε να έχουμε πολιτικές οι οποίες να συνδυάζουν την επαγγελματική ζωή ε, και ε, με την προσωπική ζωή αλλά είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Στην ουσία εδώ υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το τι σημαίνει οικογενειακή ζωή υπάρχουν κάποιες νοοτροπίες, υπάρχουν κάποιες ε, ε, διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τους γυναίκες και μερικές φορές όταν δεν υπάρχει πολλή ισότητα ε, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες βλέπουμε ότι έχουν πολλά παιδιά. Υπάρχει ένας αυξανόμενος συνεχώς αριθμός ανδρών, σαν παράδειγμα στην Ισπανία, που δεν έχει αυτή τη στιγμή οικογένεια. Άλλοι λένε όλο και περισσότερο ότι σήμερα δεν θέλουμε παιδιά, αργότερα θα δούμε, αργότερα θα κάνουμε. Ε, μέσω λοιπόν των πολιτικών ε, ε, που βοηθούν τον συνδυασμό της οικογενειακής με την προσωπική ζωή θα τους βοηθήσουμε να αποκτήσουμε. Βέβαια οι πολιτικές μέχρι τώρα δεν έχουν πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα και από την άλλη λέγουν ε, ότι θα κάνουν αργότερα παιδιά, αλλά μετά περνάει ο χρόνος, περνούν τα 40 χρόνια, ε, μειώνεται η δυνατότητα να μείνει έγκυος μια γυναίκα και υπάρχουν οριακές δυνατότητες επιστημονικές που χρησιμοποιούνται. Στον τομέα λοιπόν της γονιμότητας και ιδιαίτερα στην Ισπανία που γνωρίζω αρκετά καλά, ε, όχι μόνο οι γυναίκες ε, έχουν, υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες θέλουν λίγα παιδιά, αλλά υπάρχουν και όλο περισσότερες γυναίκες που δεν θέλουν παιδιά. βλέπουμε ότι το 50% των γυναικών που είναι σε μια ηλικία στο τέλος της αναπαραγωγικής ηλικίας στην Ισπανία έχουν κατά μέσο όρο δύο παιδιά και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που δεν έχουν καθόλου παιδί. Αυτό δεν είναι μόνο οικογενειακό θέμα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει σχέση επίσης και με τις εξωτερικές παραμέτρους. Είναι ένα περίπλοκο θέμα λοιπόν και όχι μόνο να δώσουμε κάποια κίνητρα, τα οποία σίγουρα κίνητρα είναι ε, σίγουρα απαραίτητα, αλλά το θέμα είναι πολύ πιο περίπλοκο. Είναι επίσης σημαντικό για κάποιους το να μην έχουν παιδιά, όχι μόνο στα πλαίσια αυτής, αυτού του μακροοικονομικού σεναρίου του δημογραφικού, αλλά ε, θα φτάνουν κάποιοι άνθρωποι να ζουν 100 χρόνια και να μην έχουν ε, ε, επιγόνους. Το θέμα δεν είναι μόνο ε, να ζει μόνος του για συγκεκριμένους λόγους όταν είναι θέμα επιλογής, αλλά θα αναγκάζεται σε αυτή την περίπτωση να ζήσει κάποιος πάρα πολύ μόνος του. Πρέπει λοιπόν να δούμε τη γονιμότητα περισσότερο περίπλοκα, αν θέλετε, για να καταλάβουμε για ποιο λόγο κάποιοι δεν θέλουν να έχουν παιδιά σήμερα. Νομίζω ότι οι συνάδελφοί μου απήντησαν με τόση πληρότητα που αναρωτιέμαι αν, μπορούσα, αν θα μπορούσα και εγώ κάτι να προσθέσω. Μάλλον όχι. Α, δεν θέλετε λοιπόν να προσθέσετε πορεία, Λέει καλά, ευχαριστώ πολύ. Άρα, τελειώσαμε το μέρος αυτό της ημερησίας διατάξεως. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία ε, Λοντοβίτσι καθώς και τους δύο άλλους εμπειρογνώμονες που διεύρυναν την οπτική μας για τα δημογραφικά θέματα και μας πρόσφεραν νέες ιδέες που μπορούμε να περιλάβουμε στις μελέτες μας. Ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, ελπίζω ότι δεν είναι η τελευταία επαφή σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι είτε το βλέπουμε ως πρόβλημα είτε όχι, το θέμα θα παραμείνει πάντως ενεργό για μας. Θα παραμείνει μαζί μας για πολλά χρόνια. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Και τώρα, Φρανσουά Αλφονσί, για λίγα λεπτά, γιατί ε, είμαστε αρκετά Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο το θέμα τη έκθεσή μου. Πρόκειται για έναν ευρωπαϊκό κανονισμό που θα θεσπίσει τα μέτρα τη ενία αγορά για τι ηλεκτρονικέ επικοινωνίε, ώστε να είναι μια διασυνδεδεμένη ήπειρο ε, η Ευρώπη. Γιατί αναλαμβάνεται μια τέτοια πρωτοβουλία, διότι η πρόσβαση των ιδιωτών και των επιχειρήσεων ε, στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών χωρίς περιορισμούς και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος είναι το ευκταίο και η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε αυτό το τομέα διότι είναι κατακαιρματισμένη. Έχει 28 διαφορετικέ εθνικές αγορέ με ε, ιδιαίτερότητε ε, ω προ την αδειοδότηση για την χορήγηση συχνοτήτων στη στις κανονιστικές διαδικασίες. Αυτό επηρεάζει αρνητικά τις υπηρεσίες, τη χρήση των υποδομών, τις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές και όταν ζήτε, τίθεται ζήτημα διασυνδεσιμότητας βλέπουμε ότι σε επιχειρήσεις όπως η υλικοτεχνική στήριξη, τραπεζικές υπηρεσίες κτλ. αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Ο στόχος μεταξύ άλλων είναι η αρμόνιση της αγοράς. Δεν επίπει αυτό ακριβώς στην αρμοδιότητά μας, αλλά στο μέλλον καλό θα ήταν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο στις μεθοριακές περιοχές καλό θα ήταν με τον νέο κανονισμό να εναρμονίσουμε παραδείγματο χάρη τις διαδικασίες ε, διαγωνισμών ε, για τις κρατικές προμήθειες, ε, ούτως ώστε, ε, όπως έλεγα, στις μεθοριακές περιοχές ε, να έχουμε ταυτόχρονα προσφορές από διάφορες χώρες για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Στις ψηφιακές επικοινωνίες θα τονωθεί η αγορά με τον νέο κανονισμό. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης βεβαίως έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό σε σχέση με αυτό, ε, διότι ε, αναρωτιόμαστε αν θα ε, ρυθμιστούν μόνο οι χώρες οι περιοχές με ε, πυκνό πληθυσμό ε, ή θα καλυφθούν και περιοχές που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επενδυτές. Δηλαδή η πρόσβαση ψηφιακές επικοινωνίες θα πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα καθολικής υπηρεσίας και να συνδυαστεί και μάλιστα βασικότερες υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θέλει να επενδύσει στις ευρυζωνικές. Θα πρέπει λοιπόν να συμπληρώσουμε αυτήν την πρόταση αυτή τη σύσταση, διότι ο στόχος ε, είναι να υπάρχει πανευρωπαϊκή κάλυψη ακόμη και στις νησιωτικές ε, περιοχές ε, και σε εξόγως απόκεντρες περιοχές. Στις τροπολογίες επιμένουμε για δύο ζητήματα. Γενίκευση της κάλυψης, της δυνατότητα πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες όταν αναπτύσσονται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις εκφάσεις τους και δεύτερον η εναρμόνιση ε, των εμπορικών διαδικτυακών υπηρεσιών εάν αναπτυχθούν χωρίς να ελέγχονται ε, θα υπάρξει ένας ε, κορεσμός και ο καταναλωτής θα ε, θεωρεί ότι ε, είναι υπερβολικοί ε, οι περιορισμοί που επιβάλλονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αντίθετα, οι τραπεζικές υπηρεσίες θα πρέπει να αναπτυχθούν. Οι απόκεντρες περιοχές οι υπεθρός έχουν καταναλωτές ε, που εξαρτώνται ακόμη περισσότερο από αυτές ε, τις επικοινωνίες για να συνδεθούν με τον έξω κόσμο. Λοιπόν, ε, οι χρήστες θα έχουν υπηρεσίες ακροτηριασμένες εξαιτίας της υψηλής συγκέντρωσης στις, μεγάλες, στα μεγάλα αιστικά κέντρα αυτών των νέων υπηρεσιών. Ε, τραπεζικές ε, υπηρεσίες λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες ε, τεχνολογικές δυνατότητες που μας προσφέρει το διαδίκτυο τόσο ώστε να υπάρχει ευρύτατη κάλυψη ολόκληρης επικράτησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ήθελα να σας πω και ακούω τις ερωτήσεις. Υπάρχει πρόβλημα νομίζω για τους σοσιαλιστές. Μπορείτε να μιλήσετε εσείς Γιάννη Σνίλσεν, Κωνσταντσα δεν ξέρω που είναι. Ε, ναι, ε, δεν είμαι σκιώδης. Ήθελα να κάνω μόνο κάποιες παρατηρήσεις γιατί με ενδιαφέρει το θέμα. Όταν ζει κάποιος σε αεροκατοικημένη περιοχή όπως εγώ, στη Βόρεια Σουηδία, ε, συνειδητοποιεί ότι ε, οι δυνάμεις της αγοράς ε, δεν καταφέρνουν σε τέτοιες περιοχές να δώσουν στους καταναλωτές αυτά που χρειάζονται. Δεν τα καταφέρνουν. Όταν προσπαθεί η Σουηδική κυβέρνηση να υποχρεώσει τους εμπορικούς φορείς, τους λέει πρέπει να έχουμε ευρυζωνική σε ολόκληρη τη Σουηδία. Και μας λένε όχι δεν είναι υποφελές εμπορικά, δεν ε, είναι κερδοφόρο. Άρα θα πρέπει να ασχίσουμε πίεση στους παίκτες της αγοράς. Είναι μια πολιτική επιταγή που εμείς θα τους επιβάλλουμε. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να κερδίζουν χρήματα μόνο σε περιοχές όπου ε, είναι μεγάλος ο πληθυσμός. Ε, θα πρέπει να δεχθούν και τις απώλειες ε, για τις αεροκατοικημένες περιοχές. Το άλλο που με θορυβεί είναι ότι οι μεγάλοι παίκτε ε, της αγοράς δεν κάνουν αυτό που του αναλογεί και το μόνο που του απασχολεί είναι να βγάζουν λεφτά. Ε, λοιπόν δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό και ξέρετε η ίδια κατάσταση ισχύει. Είτε μιλάμε για το εθνικό είτε για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι. Ευχαριστούμε Λάμπερτ για το Παρακαλώ. Ε, ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το θέμα είναι σημαντικό. Το διαπιστώσαμε και πριν με τα δημογραφικά. Πόσο σημαντική είναι η παροχή των υπηρεσιών αυτών και τώρα και αργότερα. Αυτό προϋποθέτει και ένα καλό δίκτυο και πρόσβαση στο δίκτυο. Ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον να καταθέσουμε της ίδιας πρωτοβουλίας. Η τεχνολογία μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά σκεφτείτε λίγο και τις νέες γενιές δορυφόρων. Κάποια, στιγμή δεν θα χρειαστεί καν να υπάρχει καλωδιακή διασύνδεση. Χρειάζονται όμως, χρειάζονται όμως χωρητικότητα και πρέπει να είναι και τεχνολογικά ουδέτερο, διότι τα πράγματα αυτά προχωρούν, οι τεχνολογίες εξελίσσονται. Δέστε τι γίνεται με την κινητή τηλεφωνία. και είναι διάφορο τώρα εάν κινείται και η κινητή τηλεφωνία μέσω διαδικτύου είτε μέσω καλωδίων. Και η συνάδελφός μου Πιλάρ Δικαστήγιο εργάζεται πάνω στην πρόταση αυτή. Πρέπει να δούμε και να αποφασίσουμε με ποιο τρόπο θα κατορθώσουμε να κάνουμε τις υπηρεσίες αυτές οικονομικότερες, φθηνότερες. Διότι μέχρι τώρα είχαν σημειωθεί και τεράστιες, τεράστια περιθώρια κέρδους μέχρι και 800%. Και εκεί χρειάστηκε κάτι να γίνει. Πρέπει να μειωθούν οι τιμές. γιατί χρειάζεται και κάποιο ανταγωνισμό και ο ανταγωνισμό αυτός θα οδηγήσει στην πτώση των τιμών. Και για την Νότια Ευρώπη ισχύει αυτό. Είδα για παράδειγμα σε διακοπές σε νότιε ε, ευρωπαϊκές χώρες πόσο υψηλέ είναι οι τιμές της χρήση του διαδικτύου. Ενώ το διαδικτύο είναι απαραίτητο και για πολύ ουσιώδεις υπηρεσίε. Πρέπει λοιπόν να δούμε και από κρατική πλευρά να υπάρξουν ρυθμίσεις που να μην επιτρέψουν τα υπερβολικά αυτά περιθώρια κέρδους. Όπως είπα αυτά πρέπει να εξεταστούν. Και να μην δημιουργηθούν συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που να μπορούν να εκμεταλλευτούν κάποια δεσπόζουσα θέση στην αγορά πρέπει να έχουν και οι μικροί πάροχοι υπηρεσιών τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Βλέπω ότι υπάρχουν ακόμη χώρες μέλη που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και που θα ήθελαν να παραμείνουν τα ολιγοπόλια αυτά. Αλλά δεν είναι αυτή η ιδέα που έχουμε εμείς για την ενιαία αγορά. Ο καθένας πρέπει να έχει πρόσβαση στην αγορά και οι επιχειρήσεις μας να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν και διαμεθοριακά και ενδεχομένως να αποκομίσουν κέρδη από τη δραστηριότητά τους αυτή. Ευχαριστώ πάντως για τη σωστή ανάπτυξη του θέματος από το συνάδελφό μου. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Ήθελα να σας πω πως... Ε, Επειδή πλησιάζει το τέλος της θητείας, θέλω να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας προσπαθήσαμε να γνωμοδοτήσουμε για όλες τις ε, συνιστώσεις ε, της πολιτικής αυτής ε, από τη δική μας σκοπιά γιατί συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη η εδαφική διάσταση και τονίσαν πόσο σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση στις υπηρεσίες στα δίκτυα σε όλα τα εδάφη της Ένωσης όσο απομακρυσμένα και αν είναι και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό Ελπίζω οι συνάδελφοι μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία για τις τροπολογίες ε, να ε, φροντίσουν ώστε να αποτυπώσουν τις ιδέες τους ε, σε τροπολογίες. Μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων επίσης μπορούμε να συμβάλλουμε στην βελτίωση της πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες της εσωτερικής αγοράς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, η ουδετερότητα του διαδικτύου που μας είπε ο Λάμπερτ είναι ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Εδώ και δεκαετίες ε, τη διακριτική μεταχείριση ε, για τις δορυφορικές υπηρεσίες η Ένωση, ενώ αυτό μπορεί να αποτελέσει την απάντηση για τις απομακρυσμένες απόκεντρες περιοχές. Ξαναλέω, ελπίζω η ΣΝΑΛΦΟΥ δεν είναι εδώ. Ε, να εκμεταλλευτούν ε, τις μέρες που μας μένουν μέχρι να εκνοήσει προθεσμία, 20 Δεκεμβρίου δηλαδή, για να καταθέσουν τροπολογίες. Εμείς θα ψηφίσουμε τον Ιανουάριο και η Επιτροπή Βιομηχανίας το Φεβρουάριο. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την καταληκτική ημερομηνία, διότι για να καταφέρουμε να φτάσουμε γρήγορα στην Ολομέλεια ε, πρέπει να τηρήσουμε αυτό το περιοριστικό χρονοδιάγραμμα. Ε, Φρανσό Αλφόνση, θα θέλετε να προσθέσετε κάτι μετά από αυτή τη σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Όχι, όχι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σημείωσα βεβαίως όλα αυτά ε, που μας είπαν οι συνάδελφοι. Δεν το γνώριζα το θέμα. Αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντικό είναι σε περιφερειακό επίπεδο, αν υπάρχουν πιο πεφωτισμένοι από μένα, να μου καταθέσουν παρακαλώ τροπολογίες ε, για να βελτιωθεί το κείμενο. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Ε, Α περάσουμε στο τελευταίο βασικό σημείο τη μέση διάταξη. Ο Νίκολα Μάρτιν είναι ήδη εδώ και μπορούμε να αρχίσουμε λίγο νωρίτερα. Αυτή είναι η φώτιση που περιμένουμε να μας έρθει από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ποιο τρόπο μπορούμε να χειριστούμε πιο αποτελεσματικά τις εκτελεστικές πράξεις και τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Ε, Νίκολας, ε, ε, όταν διακοπούν οι κοινοβουλευτικέ εργασίε εν των εκλογών, νομίζω ότι είναι σημαντικό να εντείνουμε τη συνεργασία μας, ούτω ώστε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με τις κατεξουσιότητες και τις εκτελεστικές πράξεις. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να κάνω σε 5-10 λεπτά είναι να σα δώσω μια περιγραφή των εφαρμοστικών πράξεων όπως επίσης και των κατεξουσιοδότησης πράξεων όπως προβλέπονται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε διαμορφώσει το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο όμως θα πρέπει να συμπληρωθεί με τις δευτερεύουσες πράξεις όπως σας είπα. Έχουμε δύο ειδών, τις εφαρμοστικές όπως είπα πράξεις και τις κατεξουσιοδότηση πράξεις ε, απαιτούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες για κάθε μία από αυτές. Υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται. Η κατεξουσιοδότηση πράξης είναι πράξεις οι οποίες συμπληρώνουν αν θέλετε τα μία απαραίτητα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις νομοθετικές πράξεις και η κατεξουσιοδότηση πράξης υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τίθενται σε ισχύ μετά από μια χρονική περίοδο δίμηνη εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή από πλευράς του Συμβουλίου. Οι εφαρμοστικές πράξεις από την άλλη έχουν σαν στόχο να διαμορφώνουν τις ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή της βασικής νομοθετικής πράξης. Οι εφαρμοστικές πράξεις είτε υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς την διαδικασία της επιτροπολογίας ή περνούν από την ε, επιτροπολογία μέσω της νέας επιτροπής που έχει διαμορφωθεί ε, ε, μέσω της νέας επιτροπής που διαμορφώθηκε για τα διαρθρωτικά ταμεία. Μιλάμε για δύο διαφορετικές διαδικασίες δηλαδή. Τώρα θα, συγκεντρώσω την προσοχή μου στις κατεξουσιοδότηση πράξεις όπου το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να σταματήσει τη θέση σε ισχύ αμφισβητώντας την μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ενώ για τις εφαρμοστικές πράξεις δεν έχει καμία τέτοια άμεση δυνατότητα, απλά ενημερώνεται μέσω της διαδικασίας μεταφοράς των εγγράφων ε, γνωστοποίησης καλύτερα των εγγράφων όταν ε, τα έγγραφα αυτά αποστέλλονται και στα κράτη-μέλη μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας. Ο βασικός στόχος από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο για τη νέα περίοδο είναι πλήρες πλέον ή μάλλον να συμπληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Και γι' αυτό ακριβώς προετοιμάζουμε τις πράξεις αυτές με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα για τις εφαρμοστικές πράξεις έχουμε πάντα υπόψη ότι υπάρχει ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο λόγω των διακοπών και αυτό δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Θα ήθελα λοιπόν να σας περιγράψω το χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε μια προτεραιότητα, αν θέλετε, των διαφορετικών αρμοδιοτήτων που είναι απαραίτητε για να προχωρήσουμε στις κατεξουσιοδότηση πράξη. Η πιο σημαντική από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο κώδικα συμπεριφορά στο θέμα τη εταιρική. Ε, θέλουμε να υιοθετηθεί το ταχύτερο δυνατόν και να τεθεί σε λειτουργία το ταχύτερο δυνατόν γιατί είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία για την προγραμματική περίοδο που θα ακολουθήσει. Γι' αυτό ακριβώς και σκοπεύουμε να υιοθετηθεί αυτό στις αρχές Ιανουαρίου. Θα ήθελα να πω επίσης εισαγωγικά ότι για να διασφαλίσουμε ότι τα πράγματα μπορούν να προχωρήσουν με ταχύτητα έχει ήδη προηγηθεί κάποια προεργασία. Ξεκινήσαμε νωρίς λοιπόν ε, το 2013 με ανεπίσημες συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, με εμπλοκή εκπροσώπων από τα κράτη-μέλη, έχοντας προσκαλέσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προετοιμάσουμε επίσης τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Αυτό λοιπόν η προεργασία μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με αρκετά υψηλή ταχύτητα. Αυτό ισχύει και για τον κώδικα συμπεριφοράς αλλά και για άλλους τομείς. Για τον κώδικα συμπεριφοράς ήδη έχουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, οδηγήσει σε συναντήσεις εμπειρογνώμονες έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει τη συγκεκριμένη πράξη στις 7 Ιανουαρίου. Στόχος μας είναι λοιπόν ε, η πράξη αυτή να γνωστοποιηθεί προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο την 7η Ιανουαρίου. Αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Στη συνέχεια έχουμε μια εβδομάδα αρμοδιοτήτων αν θέλετε η οποία οδηγεί στην δεύτερη κατεξουσιοδότηση πράξη. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα έγιναν συναντήσεις εμπειρογνωμόνων έτσι ώστε να εξεταστεί το περιεχόμενο της δεύτερης αυτής πράξης και να διασφαλιστεί η σωστή της προπαρασκευή. Η πράξη αυτή καλύπτει πάρα πολλά θέματα, όπως μπορείτε να δείτε στο έγγραφο το οποίο έχετε μπροστά σας Υπάρχουν εντελώς διαφορετικά θέματα που έχουν σχέση με τα χρηματοδοτικά μέσα, με το αποθεματικό επιδόσεων, με διάφορες δράσεις ε, παραγωγής πρόκλησης οδήματος ε, ε, και επίσης και τις ελεγκτικές διαδικασίες σχετικά με τις σοβαρές αδυναμίες της λεγόμενης. Είναι σημαντικά θέματα λοιπόν τα οποία συμπληρώνουν τις βασικές νομοθετικές πράξεις οι οποίες ισχύουν στον συγκεκριμένο τομέα και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα αυτά τα θέματα να έχουν ξεκαθαριστεί στην αρχή της επόμενης προγραμματικής περίοδου, κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο να έχουν καλυφθεί όλα αυτά τα θέματα στα πλαίσια λοιπόν της συγκεκριμένης μίας ε, μοναδικής ε, ε, κατεξουσιοδότηση πράξης η οποία θα πρέπει να υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα του μηνός Φεβρουαρίου. Οι δύο αυτές λοιπόν πρώτε, κατ' εξουσιοδότηση πράξη, ο κώδικας συμπεριφορά και η δεύτερη αυτή με τα πολλαπλά θέματα, θα υιοθετηθούν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο θα επιτρέψει ε, να περάσουν δύο μήνες μετά από την τελική προθεσμία, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ολοκληρωθεί τότε η διαδικασία. Στόχος είναι όλα αυτά τα θέματα να τεθούν σε λειτουργία πριν από την διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου. Έχουμε επίσης και ένα χαμηλότερο θα έλεγα επίπεδο προτεραιότητας από αυτό στο οποίο αναφέρθηκα τώρα. Απαιτείται μια κατεξουσιοδότηση πράξη σαν παράδειγμα για την αηφόρο ανάπτυξη των πόλεων, των αστικών περιοχών, ε, μία άλλη πάλι για τη διαχείριση των δράσεων, ε, πρόκειται για χαμηλής προτεραιότητας ή να το πω καλύτερα χαμηλότερης από τις προηγούμενες σκοπεύουμε να υιοθετήσουμε τις πράξεις αυτές, αν πάνε όλα καλά, αρχές Μαρτίου και θα ενημερώσουμε γέρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υιοθέτηση της συγκεκριμένης πράξης πριν από την διακοπή επαναλαμβάνω των εργασιών του Κοινοβουλίου. Και στη συνέχεια έχουμε επίσης ακόμα χαμηλότερο επίπεδο προτεραιότητας που μπορεί να περιμένει μέχρι και το δεύτερο εξάμεινο του επόμενου έτους αυτό αφορά την εταιρική σχέση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Έχουμε την εντολή, όπως επίσης και τα θέμα της, της καταγγελίας και της ανάκτησης ή της μη δυνατότητας ανάκτησης ποσών κτλ. Αυτή είναι λοιπόν η κατηγοριοποίηση την οποία εμείς καταφέραμε να διαμορφώσουμε και η οποία ελπίζω θα μας επιτρέψει τα πιο σημαντικά τα στοιχεία, από τα στοιχεία αυτά να είναι σε θέση λειτουργίας στις αρχές της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Για να συμπληρώσω λίγο το τοπίο αν θέλετε, να περάσω και στις εφαρμοστικές πράξεις. Κάποιες από τις εφαρμοστικές πράξεις δεν απαιτούν η μορφή επιτροπολογίας, αλλά παρόλα αυτά είναι σημαντικές και πρέπει να υιοθετηθούν στην αρχή της προγραμματικής περίοδου γιατί καθορίζουν σαν παράδειγμα τις επιλέξιμες περιοχές για επενδύσεις στον τομέα της απασχόλησης και ανάπτυξης και τις διαφορετικές επίσης κατανομές, όπως επίσης και τα λεγόμενα ETC. Αυτά όλα λοιπόν θα επιτρέψουν να ε, συγκεκριμενοποιηθούν από τα κράτη-μέλη οι κατηγορίες και τα ποσά για τα ETC θα υπάρξει μια επιπλέον συμπληρωματική ε, τέτοια εφαρμοστική πράξη που θα καθορίσει τα εδάφη στα οποία θα εφαρμοστούν. Αυτά όλα θα γίνουν στις αρχές του, του επομένου έτους, αλλά χωρίς την διαδικασία επιτροπολογίας, το Φλεβάρι, αρχές Φλεβάρι, το αργότερο. Έχουμε επίσης ε, και μια υψηλή προτεραιότητα εφαρμοστικών πράξεων που έχουν σχέση τον με τον προγραμματισμό. Η προτεραιότητά μας δηλαδή με επιτροπολογία είναι τα λεγόμενα πρότυπα για τα λειτουργικά προγράμματα και κάποια κομβικά στοιχεία που αφορούν θέματα όπως την εικόνα αλλαγών και την κατηγοριοποίηση και τα συστήματα κατηγοριοποίησης. Στόχος εδώ είναι να περάσουμε ε, στη νέα επιτροπή για τα ταμεία στα μέσα Ιανουαρίου. Και αν δεν τεθούν άλλα θέματα από τα κράτη-μέλη, αυτές οι εφαρμοστικές πράξεις θα πρέπει να γίνουν δεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά και από την ε, σύσταση ή την γνωμοδότηση της ειδική αυτής επιτροπής ε, στα μέσα Φεβρουαρίου. Έχουμε επίση και μια δεύτερη προτεραιότητα για άλλα θέματα, κάποια επιτέων πρότυπα, κάποιες μεθοδολογίες, σαν παράδειγμα συγκέντρωση και σόρευση δεδομένων προς αξιολόγηση κτλ. Πρόκειται για τη δεύτερη προτεραιότητα και θα ακολουθήσουν χρονικά. Αλλά ελπίζουμε μέχρι το τέλος Μαρτίου και εκεί και αυτή η συγκεκριμένη ε, πράξη εφαρμοστική να έχει γίνει δεκτή. Αυτά. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Στόχος είναι αυτή τη στιγμή υιοθετηθούν τα προγράμματα αυτά, τα κράτη-μέλη να έχουν ήδη έτοιμα το σύνολο των κανόνων που θα δημιουργηθούν από τις εφαρμοστικές πράξεις και από τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των κύριων πράξεων. Θα συνεργαστούμε φυσικά όσο μπορούμε καλύτερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις για να διασφαλίσουμε μια ομαλή διαδικασία. Θα προσπαθήσουμε επίσης να επιταχύνουμε τη θέση σε ισχύ χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν από πλευράς Κοινοβουλίου και Συμβουλίου να υποδείξουμε πριν από το τέλος της, της ε, δίμηνης περίοδου ότι δεν θα, ε, ε, δεν θα εμφανίσουν αντιρρήσεις σε σχέση με τις κατεξουσιοδότηση κυρίως πράξεις. Και μπορούμε φυσικά να περιμένουμε και από πλευρά σας περαιτέρω προτάσεις έτσι ώστε να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Ευχαριστώ Νίκολας. Σήμερα πήραμε απόφαση σαν Περιφερειακή Επιτροπή οι εισηγητές μας για τις πράξεις αυτές να είναι οι εισηγητές που ήταν στην βασική νομοθετική ρύθμιση και που γνωρίζουν τα θέματα. Το ερώτημά μου τώρα, για αυτόν τον κανόνα που είπατε στο τέλος της παρουσίασής σας, της μη παρουσίασης αντιρρήσεων, το αίτημα θα πρέπει να προέλθει πρώτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει δηλαδή να τεκμηριώσετε κατά κάποιο τρόπο το αίτημά σας προς το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να μην προβάλλουμε αντιρρήσεις και να ανταποκριθούμε θετικά. Αφού το συζητήσουμε βέβαια. Και όπως και να έχουν τα πράγματα πάντως από σας θα εξαρτηθεί χρονικά το πράγμα. Έχετε σκεφτεί σε ποιες από αυτές τις κατεξουσιοδότηση πράξεις θα μπορούσατε να ζητήσετε από το Κοινοβούλιο μία δήλωση μη κατάθεση αντίρρησης. Νομίζω ότι ιδίω για τον κώδικα δεοντολογίας, όπου νομίζω ότι υπάρχει κοινό συμφέρον των δύο οργάνων να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό. Όπως γνωρίζετε, αυτό περιλαμβάνεται ρητά, η αναδρομική του ισχύ περιλαμβάνεται ρητά στο βασικό κανονισμό. Θα είναι καλό λοιπόν να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ, όπως είπα, το δυνατό συντομότερο. Για την δεύτερη κατεξουσιοδότηση πράξη θα είναι μία ενία η οποία θα καλύπτει όλες αυτές τις εξουσιοδοτήσεις, empowerment, και ίσως είναι κάπως πιο περίπλοκο να επιταχυνθεί εκεί η διαδικασία διότι θα απαιτήσει εξέταση και από πλευράς Κοινοβουλίου και από πλευράς Συμβουλίου και ίσως εκεί υπάρχει λιγότερο περιθώριο για να μπει ταχύτερα σε ισχύ. Αλλά αυτό πάντως είναι κάτι το οποίο θα το διερευνήσουμε στο προπαρασκευαστικό στάδιο, αν υπάρχει δηλαδή ρεαλιστικά κάποια τέτοια δυνατότητα. Πρόεδρος Ιούπνερ, Λαμπέρ, μιας και ο άλλος αρμόδιος δεν είναι εδώ, θα θα μπείτε σε διαθεσμική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξετάσετε εάν είναι δυνατόν να εγκριθεί αυτή η διαδικασία μη προβολής ενστάσεως από την αρχή. Θα χρειαστεί μάλλον πολλή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων για να επιτεθεί ο σκοπός αυτός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει κιόλα να υποβάλει και τις σχετικές πληροφορίες για αυτή την Early No Objection Procedure και στο Συμβούλιο. Λαμπέρ, Λάμπερ, Μανίστερ, Ρόι, θέλετε να πείτε κάτι. Α, Γιάνν Όλμπριχτ. Ίσως να μην πρόσεξα κάτι. Αν, το, αν δεν το πρόσεξα, όντω ε, ζητώ συγγνώμη που κάνω τελικά την ερώτηση. Η διαδικασία είναι ξεκάθαρη. Αν δεν υπάρχει ένσταση. Αν υπάρχει ένσταση όμω, τότε ποια είναι η διαδικασία. Αν προβληθεί ένσταση από πλευρά μα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για αυτά, για, αυτό για μα. Ίσως να το εξήγησε, αλλά ίσως να μην το πρόσεξα. έχετε το σημείωμα αυτό που έχει ε, συντάξει η Γενική Διεύθυνση που περιλαμβάνει όλα τα βήματα. Μπορούμε να ζητήσουμε και όλα εδώ βέβαια από τη γραμματεία αντί να τα πω εγώ να τα πείτε καλύτερα εσείς. Πολύ σύντομα η διαδικασία περιλαμβάνεται ίσως όχι πολύ σαφώς μέσα στον κανονισμό. Με λίγα λόγια, από τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί στην Ολομέλεια η κατεξουσιοδότηση πράξη όπως οποιαδήποτε άλλη διαβιβαζόμενη πράξη από την Κομισιόν υπάρχει μια ε, προθεσμία δύο, δύο μηνών και μπορεί να επεκταθεί για άλλους δύο μήνες. Υπάρχει και άλλη διαδικασία που ανέφερε η Πρόεδρος που μπορεί να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν διαβιβάζει την κατεξουσιοδότηση πράξη που συνεπάγεται ότι Συμβούλιο και Κοινοβούλιο αντιδρούν πριν από το πέρας των δύο μηνών με αποδοχή. Άρα υπάρχει ανάγκη να γίνει μια ενέργεια αποδοχής της κατεξουσιοδότησης πράξης. Αν δεν αναλυθεί καμιά δράση ή αν δεν προταθεί η επίουσα διαδικασία από την Κομισιόν μετά την πάροδο των δύο μηνών και αφού έχει ανακοινωθεί στην Ολομέλεια ή στο Συμβούλιο θεωρείται τότε η κατεξιότητα πράξη ότι έχει εγκριθεί. Αν θέλουμε να δράσουμε διότι υπάρχει κάτι που δεν μας αρέσει ή θέλουμε να ανακληθεί η ανάθεση αρμοδιοτήτων, τότε προβλέπεται διαδικασία στον κανονισμό που οδηγεί στην έγκριση από το Κοινοβούλιο προτάσεως ψηφίσματος που ενδέχεται να κάνει συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει το α ή το β ή μπορεί να φτάσει και μέχρι την ανάκριση της κατεξουσιοδότηση αρμοδιότητας. Άρα πρόταση ψηφίσματος που συντάσσεται από τον εισηγητή συζητείται σε κοινοβουλευτική επιτροπή, εγκρίνεται σε κοινοβουλευτική επιτροπή και διαβάζεται στην Ολομέλεια, όπως οποιαδήποτε άλλη έκθεση. Αυτή με λίγα λόγια είναι η διαδικασία που έχει ίσως και κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες εδώ και εκεί, αλλά περίπου αυτό είναι. Η πρόεδρος Ντανούτα. Για την περίπτωση της κατεξουσιοδότησης πράξης μπορούμε εμείς να προβάλλουμε ένσταση για οποιονδήποτε λόγο. Όλμπριχτ στο συγκεκριμένο αυτό έτος θα είναι περίπλοκα τα πράγματα. Αν δεν υπάρχουν στάσει, έχει καλώς. Εκτός από την Delegated Act υπαριθμών 4 που θα πάει τον Ιούλιο με το νέο κοινοβούλιο. Ενώ η 1 έως 3 θα πάνε στο παλιό κοινοβούλιο. Και βέβαια η τελευταία ολομέλεια του κοινοβουλίου, του τρέχοντος κοινοβουλίου είναι τον Απρίλιο. Αν λοιπόν λάβουμε κάτι τον Μάρτιο Εάν δεν υπάρχουν στάσεις έχει καλώς. Αν όμως υπάρχει λόγος ένστασης τότε όλη η διαδικασία θα πάει στο επόμενο κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί. Ναι, Γιάννη πρόσεξε. Θεωρητικά η Κομισιόν μπορεί να διαβιβάσει τις πράξεις αυτές μέχρι τον Μάρτιο. Αλλά για να εγκριθούν με τη συνήθεια διαδικασία αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον τις διαβιβάσουν μέχρι μέσα Φεβρουαρίου. Μα εδώ μιλάμε για, Φεβρου... για Μάρτιο. Εδώ λέει Μάρτιο στο χαρτί. για όσα διαβάσετε τον Μάρτιο δεν γίνεται πλέον η συνήθη διαδικασία που παίρνει δύο μήνες γιατί η τελευταία ολομέλεια είναι τον Απρίλιο. Γι' αυτό είχα θεωρήσει ότι οι τελευταίες πράξεις που μπορεί να σταλούν θα πρέπει να είναι μέσα Φεβρουαρίου. Ε, ναι, αλλιώς θα πάνε τον Ιούλιο, δεν ναι, Μικέλ. έγιναν διαθεσμικές συζητήσεις μεταξύ των τριών θεσμών και είπαν ότι το αργότερο 13 Μαρτίου θα είναι η τελευταία ε, προθεσμία ανακοίνωση στην Ολομέλεια ε, μιας ε, κατεξίωσης πράξης που δίνει, που δίνει μπορούμε να προβάλλουμε ένσταση τον Απρίλιο. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι αν έχουμε επιφυλάξεις και τις υποβάλλουμε στην τελευταία ολομέλεια με πρόταση ψηφίσματος, εάν αυτή η πρόταση ψηφίσματος η ε, προβάλληση στάσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να τις δεχτεί και να επανέλθει. Ιωάχιμ Τέλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στον κανονισμό μόνο στο 17α ε, αναφέρονται σε κατεξιότητα πράξη. Στο χρονοδιάγραμμα όμως δεν εμφανίζεται καθόλου, ούτε καν μέχρι το καλοκαίρι του επομένου έτους. Κάτι που δεν κατανοώ. Μιλούμε εδώ για ένα κανονισμό περιορισμένου εύρους. Θα έπρεπε να είναι δυνατόν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει κάτι για αυτήν την κατεξουσιώτηση πράξη έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσα στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία να αποφασίσουμε. Άλλες ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Νίκολα, σας παρακαλώ. Ε, κυρίως για να απαντήσετε στον Γιώαχιμ Ζέλερ. Ευχαριστώ για το τελευταίο σημείο που αφορά το EGTC, τον κανονισμό. Πρόθεση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρουσιάσουμε ένα νέο κατάλογο που να παρουσιάζει και το EPTC. Αλλά εν πάση περιπτώσει η συγκεκριμένη κατεξουσιοδότηση πράξη αφορά τους δείκτες για την αξιολόγηση και αναφορά και γι' αυτό τον λόγο δεν είναι βασική προτεραιότητα, ε, δεν πρέπει σε αυτή τη φάση να γίνει κάτι. Και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα χρόνου που έχουμε θα μπορούσαμε να το αφήσουμε σε χαμηλό βαθμό προτεραιότητας. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι κάτι άμεσο στην παρούσα φάση. Πρόθεσή μας είναι τέτοιου είδους θέματα να απασχολήσουν το νέο κοινοβούλιο μετά το καλοκαίρι. Για τα υπόλοιπα θέματα, όπως είπε ο Μιγγέλ, πράγματι θα υπάρξει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, αυτή τη στιγμή η διοργανική συμφωνία πάρει την τελική της μορφή. Αυτός είναι ο στόχος και θα υπάρξουν ίσως κάποιες αλλαγές για να προσαρμοστούμε. Αλλά οι πρώτες τρεις καταξιοδότηση πράξεις στις οποίες αναφέρθηκα θα πρέπει να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν εφόσον δεν υπάρχει ένσταση αντίρρηση από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου ε, θα μπορέσουν να τεθούν σε ισχύ. Κατανοούμε ότι στην περίπτωση που υπάρξει ένσταση, τότε σε αυτή την περίπτωση η κατεξουδότηση πράξη σε αυτη την περιπτωση η κατεξιοδοτηση πραξη απλα δεν θα τεθεί σε ισχύ. Υπάρχουν διάφορες επιλογές από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, μία επιλογή είναι να προετοιμάσει μια νέα εφαρμοστική πράξη, μια νέα κατεξιοδότηση συγγνώμη πράξη, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα θέματα που δημιούργησαν την αντίρρηση, για να μην υπάρξει εκ νέου μια τέτοια ένσταση. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θα περάσει στο νέο κοινοβούλιο αν συμβεί κάτι τέτοιο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές του 2014. Αυτό θα είναι πρόβλημα γιατί έχουμε συγκεκριμένες εντολές, αρμοδιότητες πλέον οι οποίες θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο να βρούμε κάποια τελικά κείμενα νωρίτερα. Ελπίζω λοιπόν μετά από επαφές τους επόμενους μήνες να μειώσουμε τους κινδύνους που θα μπορούσαν να θέσουν σε αμφισβήτηση ε, τις συγκεκριμένες αυτές κατεξιοδότηση πράξεις. Η κατεπίγουσα διαδικασία επιτρέπει την άμεση δημοσίευση και τέση σε ισχύ ε, μιας ε, ε, κατεξιότητας πράξη. Αλλά δεν προβλέπεται στον κανονισμό και δεν είναι κάτι το εφαρμόσιμο. Η άλλη δυνατότητα η οποία προβλέπεται είναι η πρόορη έγκριση όπου το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να δηλώσουν σκόπιμα ότι δεν θα γύρουν ενστάσεις. Ε, ενωρίτερα στη διαδικασία δηλαδή θα δηλώσουν ότι δεν θα υπάρξουν τέτοιου είδους ενστάσεις. Και όπως είπα, ιδιαίτερα για τον κώδικα συμπεριφοράς και την εξαρτώμενη από αυτό κατεξοριότηση πράξη, αυτό είναι κάτι το οποίο θα δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό βέβαια θα ισχύσει μόνο εφόσον και τα δύο όργανα είναι διατεθειμένα να συμβάλλουν. Ευχαριστώ, δεν υπάρχουν άλλα σχόλια γύρω από τα θέματα που ακούσαμε από τον Νίκολα Μάτιν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναλάβαμε την υποχρέωση και από τις δύο πλευρές να συνεργαστούμε επί των πράξεων αυτών. Θα ήθελα επίσης να πω ότι το τελευταίο είναι οι αποφάσεις τις οποίες έλαβαν οι συντονιστές. Σε περίπτωση που υπάρξει και άλλη έκθεση ιδίας πρωτοβουλία από την Επιτροπή Προϋπολογισμών επί το οποίο προς το παρόν δεν υπάρχει έγκριση από πλευρά στη διάσκεψη των Πρόεδρων σε περίπτωση που εγκριθεί το ΕΛΚΑ και οι φιλελεύθεροι αποφασίσουν ποια ομάδα τελικά θα αναλάβει αυτή την έκθεση για τις εκτελεστικές και τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Αποφασίσαμε ότι για το βασικό, οι εισηγητές του βασικού κανονισμού κάθε φορά θα είναι οι συγγητές και για αυτές τις πράξεις, για τις δημόσιες ακροάσεις. Οι συντονιστές πρότειναν ενδεχομένω να διεξαχθεί ε, και άλλη μια ακρόαση για τις ε, συμβάσεις, ε, για τις συμπράξεις σε δημόσιο ιδιωτικού τομέα. Οι συντονιστές θα επεξεργαστούν τις που θα υποβάλουμε στη διάσκεψη των Προέδρων. Γι' αυτό. Αυτά. Η επόμενη συνεδρίαση, ένα λεπτό, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, θα γίνει στις 22 και 23 Ιανουαρίου. Υπό τα διάφορα δεν έχουμε τίποτε άλλο, ούτε για κανείς άλλος. Δεν, δεν έχει ζητήσει Α, ναι. Θα γίνει ένα κοκτέιλ εδώ απ' έξω ε, στις Έξι βεβαίως, όχι τώρα, οπότε δεν ξέρω αν θα ξαναεπιστρέψει κάποιο σε μισή ώρα από τώρα, σε 20 λεπτά μάλλον από τώρα. Υπάρχουν πολλά κοκτέιλ, τέλο πάντων θα γίνει και εδώ ένα, όχι στι 6.30, στι 6. Καλά Χριστούγεννα σε όλου. ευτυχισμένο το καινούριο έτος και θα τα πούμε στο κοκτέιλ εδώ απ' έξω.